Good afternoon, lady. Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Θερμά ευχαριστώ όσους ε, ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης. Φαντάζομαι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα καταφτάσουν στην πορεία. Έχετε ήδη λάβει την ημερήσια μας διάταξη και πριν την εγκρίνουμε ε, θα ήθελα να καταγράψουμε και επισήμως την βαθιά μας θλίψη για το θάνατο ενός μέλους της Επιτροπής του κυρίου Γιάνς Νίλσον, που απεβίωσε στις 13 Μαρτίου. Ήταν 61 ετών. Ε, αφού διτέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Östersund στη Σουηδία, ο κύριος Νίλσον εξελέγει ευρωβουλευτής το 2011 και επανεξελέγει το 2014 ήταν μέλος ε, της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ήταν επίσης μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κάτι που δείχνει την προσήλωσή του στην εκπροσώπηση των ε, συμφερόντων των περιφερειών, που είναι μακριά και από τις πρωτεύουσες. Ήταν πολύ καλός συνάδελφος ε, και πολύ αξιόλογος άνθρωπος, θα μας λείψει πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να γερθούμε και να τηρήσουμε ενό λεπτού σιγή σε ένδειξη σεβασμού προς τον κύριο στο θάνατο του κύριου Νίλσον. Thank Σας ευχαριστώ και να περάσουμε στα δικά μας. Καταρχήν μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, μήπως υπάρχουν απορίες ή παρατηρήσεις. Δεν βλέπω, οπότε μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης και ε, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Ιανουαρίου και των δύο συνεδριάσεων του Φεβρουαρίου. Έχει, υπάρχουν και στο διαδίκτυο τα πρακτικά, το σχέδιο πρακτικών, οπότε αν δεν υποβληθούν ε, παρατηρήσεις ε, μέχρι το τέλος συνεδρίας θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα. Επόμενο σημείο, ανακοινώσει της Προέδρου. Να σας ενημερώσω ότι στις 9 Μαρτίου έλαβα μέρος σε μία συνεδρίαση που οργάνωσε η Βουλγαρική Προεδρία στη Σόφια με θέμα το μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών, κυρίως Υπουργοί Οικονομικών των χωρών μελών και επίσης ο πρόεδρος Επιτροπής των Περιφερειών, ο κ. Λάμπερτς, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου κ. Σιλένε, καθώς και ο Επίτροπος Φέτιγκερ. Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ο συνάδελφος Γιάν Όλμπριχτ παρουσίασε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και υποφαινομένη παρουσίασε την θέση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για το μελλοντικό ΠΔΠ βάσει της γνωμοδότησης που εγκρίναμε στην Επιτροπή μας. Όπως είπα, η συζήτηση ήταν πολύ ανοιχτή και ενδιαφέρουσα και ακούσαμε τις απόψεις ε, των κρατών μελών, διαπιστώνοντα τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του και τις δυσκολίες ό,τι αφορά τη διαμόρφωση μιας ενιαίας θέση του Συμβουλίου για το μελλοντικό πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Επίτροπος ε, Τίνκερ μας έδωσε πολύ λίγα στοιχεία, οπότε Περιμένουμε ακόμη την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το μελλοντικό ΠΔΠ που αναμένεται να δημοσιευτεί στις 2 τρέχοντος Μάιου. Δεν βλέπω κανέναν αντιπρόεδρο, οπότε το θέμα της ενημέρωσης ε, της αποστολής στη Βόρεια Ιρλανδία αναβάλλεται είτε για αύριο είτε για επόμενη συνεδρίαση. Παίρναμε στο επόμενο σημείο της σας διάταξης, την εξέταση της έκθεσης με θέμα την πολιτική συνοχή και την κυκλική οικονομία. Η συγητής μας είναι ο κύριος Ντάβορ Σκρλετς, που θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του. Και χωρίς άλλη χρονοτριβή θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Σκρλετς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, τα κροατικά. Και να ευχαριστήσω εκ των προτέρων του συναδέλφου που θα φορέσουν τα ακουστικά, τα τους. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης ε, που έχετε λάβει διευκολύθηκε κατά πολύ από τις άριθμες προτάσεις ε, και συστάσεις ε, που προέκυψαν στη συζήτηση της 24ης Ιανουαρίου. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση και στην ανταλλαγή απόψεων που οδήγησε στην υποβολή αυτού του σχεδίου έκθεσης. Στη συζήτηση καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η κυκλική οικονομία είναι εξαιρετική ευκαιρία για τη μετάβαση της οικονομίας μας σε ένα φιλοπεριβαλλοντικό κυκλικό μοντέλο οικονομίας που θα εδράζεται στην αηφόρο ανάπτυξη και θα επιτρέπει και την υλοποίηση των κλιματικών μας στόχων, των στόχων της διαφύλαξης των πόρων μας, των θέσεων απασχόλησης και της ε, ανταγωνιστικότητας, του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εν ώψη της, ε, των αξανόμενων απαιτήσεων της παγκοσμιοποίησης. Η κυκλική οικονομία θα μας επιτρέψει να διαφυλάξουμε τα, τις πρώτες ύλες και τα υλικά μας εντός της οικονομίας και θα, να περιορίσουμε τη δημιουργία απορριμμάτων και αποβλήτων έχουμε περίπου 8 δισεκατομμύρια τόνους ε, υλικά που μετατρέπονται σε ενέργεια ή προϊόντα και μόνο, μόνο 6% των, υλικών, των, των υλικών, 6% των υλικών αυτών, 0,6 μάλλον τόνοι δημιουργούνται από ε, ανακυκλωμένα ε, τέτοια απόβλητα. Τα περισσότερα απόβλητα δυστυχώς χάνονται στη διάρκεια της ανακύκλωσης και δεν ανακτώνται. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε, ε, να δράξουμε αυτή την ευκαιρία και ένα μεγάλο τμήμα αυτών των αποβλήτων να τα μετατρέψουμε σε ανάκτηση προϊόντων. Η σημαντικό είναι ο οικολογικό σχεδιασμό, η βιοοικονομία, ώστε να αποφύγουμε την κατασπατάληση των αποβλήτων και να τα δημιουργήσουμε, να τα μετατρέψουμε σε δευτερογενεί πρώτε ύλε στην περαιτέρω διαδικασία. Με τις ε, προτάσεις αυτές ε, θα μπορέσουμε να θέσουμε τα θεμέλια για την καλύτερη αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας. Επίσης, ε, πολλοί στόχοι άμεσα ή έμεσα μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση τη κυκλική οικονομία. Στην έκθεσή μου έχω τρία μέρη. Καταρχήν κάνω μια διάγνωση της παρούσας κατάστασης, τη ε, πολιτική συνοχή και το δυναμικό που μπορεί να, της πολιτικής συνοχής που μπορεί να επιτρέψει την ε, υλοποίηση της ε, κυκλικής οικονομίας. Στη στο δεύτερο σκέλος μιλώ για τους τομείς και το δυναμικό της πολιτικής συνοχής που μπορεί περαιτέρω να ενισχύσει την κυκλική οικονομία και την υλοποίηση των δημόσιων στόχων μας. Και στο τρίτο σκέλος της έκθεσης μιλώ για το μέλλον και προτείνω κάποιους ε, τρόπους ώστε η πολιτική συνοχή να μετατραπεί σε δημόσια πολιτική που θα επιτρέπει την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας και την υλοποίηση των στόχων της. Η κυκλική οικονομία ως νέος τρόπος των ε, οικονομικών αλλαγών θα πρέπει να γίνει δημόσια πολιτική ε, γιατί δυστυχώς το ε, τρέχον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν την αναφέρει αρκετά ώστε να επιτρέψει να υλοποιήσει τους στόχους της η πολιτική συνοχή Αφενό και η κυκλική οικονομία ΦΕΔΑΡΟΥ. Γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφιερώσει τα απαραίτητα κονδύλια και τις πρωτοβουλίες για να ε, ενισχυθεί η κυκλική οικονομία και να υλοποιηθούν οι άμεση και έμεση στόχοι της. Επίσης, θα πρέπει να αναδείξουμε το μεγάλο δυναμικό των επιχειρησιακών προγραμμάτων ε, και θα πρέπει μέσω αυτών τα κράτη-μέλη να ενισχύουν την κυκλική οικονομία ακόμη και στο τρέχον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες αναγνώρισαν την σημαντική ε, κυκλική, το, την σημασία της κυκλικής οικονομίας μέχρι της έξυπνης εξειδίκευσης και των ε, μέτρων που θα μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της πολιτικής. Επίσης, θα πρέπει οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν το δυναμικό της κυκλικής οικονομίας και να πραγματοποιήσουν ένα τεχνολογικό άλμα, ώστε να διορθώσουν τα λάθη του παρελθόντος, ε, αντλώντας διδάγματα από την εμπειρία άλλων περιφερειών. Επίσης, ε, στα συμπεράσματα μιλώ για τις ε, σημασίες των υποδομών σε ό,τι αφορά την ε, αξιοποίηση των αποβλήτων ή την αποτέφρωση, ώστε να περιοριστούν τα έξοδα από την διαχείριση των αποβλήτων. Επίση, θα πρέπει να ενισχύσουμε τι διοικητικέ ικανότητε σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Με την ενίσχυση όλων των επιπέδων, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ιεράρχηση των αποβλήτων και φυσικά να ληφθούν οι απαραίτητες ε, ε, δημόσιες αποφάσεις ε, και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το δυναμικό των πράσινων δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών και θα μπορέσουν να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για τις επενδύσεις στην κυκλική οικονομία. Έχουμε πολλές ευκαιρίες ε, με συνεργασία και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία, νέες πράσινες θέσεις απασχόλησης και ε, νέες αγορές για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες επίσης ε, να εφαρμόσουμε καλύτερα τους στόχους της κυκλικής οικονομίας και ε, πιο ορθολογική διαχείριση των κονδυλίων. Θα πρέπει τα κοινοτικά κονδύλια να χρησιμοποιούνται για το, την υλοποίηση των κοινών στόχων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το βιωτικό επίπεδο και την καθημερινότητα των πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, ε, θα πρέπει η στρατηγική για την κυκλική οικονομία να λαμβάνουν υπόψη και στα εθνικά σχέδια και στρατηγικές και επίσης να δημιουργηθεί δημόσια συζήτηση για το τρέχον και το μελλοντικό δυναμικό της κυκλικής οικονομίας, ώστε να την ενισχύσουμε όσο μπορούμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και περιμένω ήδη με ανυπομονησία τις προτάσεις σας και την συζήτηση μεταξύ μας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα οι σκιώδες εισηγητές. Ο κ. Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνει το λόγο. Καταρχάς, να σας συγχαρώ, κύριε εισηγητά, που προετοιμάσατε αυτή την έκθεση. Πιστεύω ότι έχετε συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία της κυκλικής οικονομίας. Τονίσατε πόσο σημαντική είναι η πολιτική συνοχής επίσης προς αυτό σκοπό, για την κυκλική οικονομία δηλαδή. είναι ένας τρόπος για την ανάπτυξη του μέλλοντος. Θα πρέπει να υλοποιηθεί, είναι καθήκον να την υλοποιήσουμε αυτή, αυτού του είδους την ανάπτυξη. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης, νέες ευκαιρίες και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής που μας πιέζει όλο και περισσότερο. Πριν από κανένα δύο χρόνια ήταν αδύνατον να εφαρμόσουμε μια τέτοια φιλοσοφία που να συνδέεται με την κυκλική οικονομία, αλλά τώρα άλλαξε νοοτροπία και έχουμε διάφορα πακέτα νομοθετικά, τα οποία συνδέονται ακριβώς με αυτό το θέμα. Ο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών είναι εξαιρετικά σημαντικός και επομένω πιστεύω ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία στο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι τοπικέ και περιφερειακές αρχές. Όλοι ξέρουμε ότι η εφαρμογή όλων των πολιτικών γίνεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Όπως αναφέρει και η ίδια η έκθεση, οι μεμονωμένες χώρες έχουν τη δική τους εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία. Η πολιτική συνοχής έχει θετική επίπτωση σε διάφορους άλλους τομείς. Ο εισηγητής ε, τους ανέφερε διαχείριση των αποβλήτων. Θα προσθέσω και τον τομέα της γεωργίας. Εντός της γεωργίας Έχουμε μια βιομηχανία που βασίζεται στην βιολογική χρήση προϊόντων ή στα βιολογικά προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη γεωργία. Αυτό χρηματοδοτείται με πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Χρησιμοποιούμε φυσικά υλικά, τα οποία θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα ορυκτέλια στο μέλλον. Και ορυκτά καύσιμα. Επίση, δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην δασοκομεία στην, στα πλαίσια τη εσωτερική της κυκλικής οικονομίας και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο ω κατασκευαστικό υλικό. Φυσικά τα δάση είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τη μείωση του, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και ξέρουμε ε, επίση ότι η βιομάζα είναι μια πολύ σημαντική ανέωσιμη πηγή ενέργεια. Εντό τη πολιτική συνοχή έχουμε τονίσει την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας Είμαι Σλοβαίνος και πρέπει να σας πω ότι πολλά κτίρια στη Σλοβενία έχουν ανακαινιστεί με τη βοήθεια και τα χρήματα της ε, πολιτικής συνοχής και τώρα τα κτίρια αυτά είναι πολύ πιο αποδοτικά ενεργειακά. Σε εθνικό επίπεδο ενθαρρύνουμε τις περιφέρειες, τους δήμους και τις κοινότητες να αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο τέλος της έκθεσης διαβάζουμε για το ρόλο των πόλεων στην κυκλική οικονομία. Φυσικά θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες για να τονίσουμε περισσότερο το ρόλο των περιφερειών και των περιοχών της υπαίθρου. Γιατί η περισσότερη βιομάζα παράγεται και χρησιμοποιείται στις περιοχές της υπαίθρου. Τα ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και άλλα εργαλεία που συνδέονται με την κυκλική οικονομία τα έχουμε ενσωματώσει όλα αυτά σε ένα συνεκτικό όλο. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέε πράσινε θέσει απασχόληση στην Ήπεθρο και να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε τι περιοχέ τη Ήπεθρου να κρατήσουν του κατοίκου και να σταματήσει η απερίμωση, να σταματήσει η έξοδος προς τις αστικές περιοχές γενικά. Σας συγχαίρω ακόμα μια φορά για την έκθεση αυτή και όπως σας είπα θα υποβάλω και κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάλκοβα είναι η επόμενη σκιώδηση Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω από εκεί που τελείωσαν οι προλαλήσαντες. Οι προλαλήσαντες. Ευχαριστώ την, τον εισηγητή για αυτό το κείμενο. Είναι καλή βάση για συζήτηση. Και εγώ είμαι πεπισμένη ότι η μετάβαση στην κυκλική οικονομία είναι μια τεράστια ευκαιρία για την τοπική αυτοδιοίκηση τα επόμενα χρόνια, για τους Δήμους και τους κοινότητες. Θα πρέπει λοιπόν να τα εφαρμόσουμε αυτά χάρη σε μια καλή νομοθεσία. Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία θα πρέπει να υποστηριχθεί εκεί όπου εφαρμόζεται, δηλαδή στη, στο, να υποστηρίξουμε δηλαδή, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και οπωσδήποτε να τις εμπλέξουμε. Ξέρω διάφορα παραδείγματα όπου μικρές κοινότητες, μικροί δήμοι έχουν τη δική τους στρατηγική και τελικά ανεξαρτητοποιήθηκαν σε ό,τι αφορά την, τις ενεργειακές τους ανάγκες. Η τεχνογνωσία και η γνώση λειτουργεί. Αυτό σημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να εμπλακεί στο σχεδιασμό αυτής της στρατηγικής. Και θα πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης των δικών του στρατηγικών αυτών των δήμων και κοινοτήτων στο βαθμό που θέλουν να εφαρμόσουν την κυκλική οικονομία. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνούμε την ε, ενεργειακή ανεξαρτησία και την ενεργειακή βιωσιμότητα και αποδοτικότητα σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να μπορούν να παράγουν ενέργεια και θέρμανση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα απόβλητα των ε, Δήμων και Κοινοτήτων μπορούν να τα επεξεργαζόμαστε σε σταθμούς ε, και να παράγουμε βιοαέριο ε, και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε, μπορούμε επίσης να έχουμε και σε τοπικό επίπεδο λιπάσματα. Ε, στην Ανατολική Σλοβακία ε, έχω δει ορισμένους σταθμούς βιοαερίου όπου βλέπω πώς μπορεί να βοηθήσουν αυτοί οι σταθμοί να διατηρήσουμε την παραγωγή. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η υποστήριξη μπορεί να δημιουργήσει και θέσεις απασχόλησης. Η σημερινή γραμμική οικονομία παράγει Επίσης, πάρα πολλά πλαστικά. Υπάρχουν νησιά από πλαστικά στον ωκεανό, στους ωκεανούς. Η πολιτική συνοχής, η μελλοντική πολιτική συνοχής θα πρέπει να βασίζεται σε διάφορα επίπεδα κινήτρων για να μειώσουμε τα πλαστικά απόβλητα. Και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και την ανακύκλωση, γιατί ξέρουμε ότι πολλές χώρες στην Ένωση χρησιμοποιούν ακόμα τις χωματερές και θάβουν τα πλαστικά τους. Όταν μιλάμε για την ανακύκλωση επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα κλωστεφοντουργικά, το γυαλί, το, τα κατασκευαστικά υλικά. Δεν περιοριζόμαστε κατά ανάγκη στα πλαστικά, πρέπει να έχουμε υπόψη μας και άλλα υλικά. Επίσης υποστηρίζω την ιδέα ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την κυκλική οικονομία μεταξύ των στόχων της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Γιατί πολλά από τα μέτρα που χρηματοδοτεί η πολιτική συνοχής συνδέονται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Το οποίο σημαίνει ότι αν θέλουμε να εφαρμοστεί πραγματικά αυτή η ιστορία, θα πρέπει να βοηθηθούμε και από την πολιτική συνοχή που έχει και σαφείς ορισμούς και προσδιορίζει σωστά αυτούς τους στόχους. Περιμένω λοιπόν να υποβάλουμε κάποιες, θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε και είμαι σίγουρη θα συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Τόμασιτς. Η κυρία Τόμασιτς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τρόπος α, α, απασχόλησης αλλά και γενικώ ο τρόπος ζωής που στόχο έχει την προμήθεια, γρήγορη παρασκευή και απόρριψη ε, των υλικών δεν είναι καλό μοντέλο. Γι' αυτό συμφωνώ ότι ένα τέτοιο μοντέλο παραγωγής έχει πλέον ξεπεραστεί και δεν έχει κανένα μέλλον. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση στα τέλη του περασμένου έτους υιοθέτησε το πακέτο μέτρων για την κυκλική οικονομία και μάλιστα ανήγγειλε επενδύσει 24 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επιχειρηματικά σχέδια που θα περιστρέφονται γύρω από το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Σίγουρα το μοντέλο αυτό δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις ε, στα κράτη-μέλη γιατί θα θα υποχρεώνει σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές. Αλλά χωρίς ε, καλά σχεδιασμένη πολιτική δεν πρόκειται να ευοδοθεί η κυκλική οικονομία. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε τα πρότυπα, τις προδιαγραφές, τους στόχους και να παρακολουθούμε την εφαρμογή τους. Ε, όπως πολύ σωστά είπε ο εισηγητής, υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της κυκλικής οικονομίας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως ε, το σύστημα ε, αντισταθμιστικών αποζημίωσεων που δίνει ενάυσματα για την πιο ορθολογική χρήση, την ανακύκλωση, και επίσης ε, τον περιορισμό των δαπανών ε, και την κατάργηση των μίας χρήσης ε, συσκευασιών. Θα πρέπει να βρούμε πιο βιώσιμες λύσεις, γιατί σίγουρα θα πρέπει να προωθούμε και την καινοτομία στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, χάρη στην κυκλική οικονομία. Επίσης θα πρέπει να δίνουμε κίνητρα στους καταναλωτές να αλλάξουν την καταναλωτική του συμπεριφορά και την συμπεριφορά τους απέναντι στην κατανάλωση και να περιορίζουν τον αριθμό των απορριμμάτων ή να αγοράζουν λιγότερα για να αποφύγουμε και τη σπατάλη. Επίσης να λιπασματοποιούν τα, περισσότερο τα απορριμματά τους. Ε, επίσης να γίνεται σωστή διαλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων και να δώσουμε ενάψματα για να καταργηθούν οι μίας χρήσης συσκευασίες. Έτσι πιστεύω θα περιορίσουμε και τα αέρα του θερμοκηπίου συμβάλλοντας ε, στην ε, στον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει να το συνδέσουμε βέβαια αυτό με τα κονδύλια της συνοχής και τον ορίζοντα 2020. Βέβαια οι προτεραιότητες αλλάζουν. Μέχρι στιγμής ε, είτε δίναμε έμφαση στη διάθεση των αποβλήτων, είτε στην αποτέφρωση. Ενώ στο μέλλον θα πρέπει περισσότερο να δίνουμε ναύσματα για την λιπασματοποίηση ή την αξιοποίηση, την ανακύκλωση, ώστε να καταφέρουμε χάρη στη δευτερογενή παραγωγή πρώτων υλικών να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιακόφτσης που είναι επίσης και ο δισηγητής. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να λάβω μέρος στη συζήτηση εκπροσωπώντας τον κύριο Αουστρεβίτσιους που δυστυχώς κολλείται σήμερα και μου ανέθεσε να παρουσιάσω τις απόψεις του. επί της εκθέσεως του κυρίου Σκερλέτς. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα φυσικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή, γιατί είναι πραγματικά αξιόλογη αυτή η έκθεση και θα εντοπίσει πολύ σημαντικά σημεία για την κυκλική οικονομία και νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογα και εύστοχα τα σχόλια του εισηγητού. Θα ήθελα να πω όμως ότι η ομάδα των φιλελευθέρων στη στηρίζει πλήρως αυτό το δρόμο. Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση κατά τη γνώμη μας. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία. Γι' αυτό τη στηρίζουμε αμέριστα και στην ομάδα των φιλελευθέρων. Η σημερινή οικονομία έχει μια σειρά πόρων, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και πολλά προβλήματα με τη διαχείριση αυτών των πόρων και με τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Πιστεύω ότι τα απόβλητα, τα απορρίμματα μπορεί να γίνουν σημαντικός πόρος στο μέλλον με τη σωστή ε, αξιοποίηση. Αντί να ανακυκλώνουμε στην Κίνα τα απόβλητά μας, θα μπορούσαμε να τα αξιοποιούμε καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είμαστε έξυπνοι, αν αντιδράσουμε αμέσως στις αλλαγές, θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε τα απόβλητα σε πόρο, σε φυσικό πόρο, το ο οποίος θα συμβάλλει και αυτό στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Επίσης θα ήθελα να τονίσουμε ιδιαίτερα την ανάγκη σύμπραξης ε, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου με συμμετοχή και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ε, έχουν και αυτές τα δικά τους συμφέροντα και θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια πρόθεσης κυκλικής οικονομίας. Φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την πολιτική συνοχή σε όλα αυτά. Γιατί παρά τις ε, αντιφάσεις που μερικές φορές και τον επίμαχο χαρακτήρα του θέματος ε, των ΧΙΤΑ, πιστεύω ότι ε, θα πρέπει και η πολιτική συνοχή να συμμετέχει στο θέμα της διάθεσης των αποβλήτων. Και σίγουρα η περιφερειακή το περιφερειακό επίπεδο είναι το κατάλληλο επίπεδο για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας. Γιατί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο γίνεται η καλύτερη αξιοποίηση τέτοιων πόρων όπως μπορούν να γίνουν τα απόβλητα, να μετατραπούν δηλαδή σε πόρους. Κάτι άλλο που θα θέλαμε να συμπεριληφθεί στην έκθεση είναι η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα. Θα ήθελα πιο σοβαρά και πιο εκτεταμένα να αναπτύξουμε αυτό το σημείο που απλώς ακροθυγός το αναφέρει ο Ντάβορ στην έκθεσή του Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια βήματα εδώ στο θέμα αυτό και να συμπεριλάβουμε και άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Για παράδειγμα, τη συμμετοχή των επενδυτικών τραπεζών. Έτσι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την οικονομία μας για να κάνει πιο εύκολα τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία. Θα ήθελα εκατακλείδη να πω ότι πιστεύω πως μέσω της πολιτικής συνοχής ε, να τονίσουμε τη σημασία που έχει το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, γιατί σε κεντρικό επίπεδο δεν μπορεί μια χώρα να λύσει το πρόβλημα. Θα πρέπει η στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ ε, να υλοποιηθούν τα σχέδια. Και γνωρίζω από συμμετοχή στην ε, περιοχή της Ίστριας ε, στα Δημοτικά Συμβούλια πόσο σημαντική είναι η συμπερίληψη του περιφερειακού και τοπικού, τοπικού επίπεδου στη διαχείριση των αποβλήτων. Έτσι πιστεύω μπορούν οι περιφέρειες να συμβάλλουν στην αποτελεσματική μετάβαση προς την κυκλική οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλους κοιόδους εισηγητές. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Η κυρία Νταμάτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ αντικαθιστώ την κυρία Αντινόρφη, η οποία δεν μπορούσε να έρθει. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε το πακέτο μέτρων για την κυκλική οικονομία για να βοηθήσει τις ε, ε, επιχειρήσεις και τους Ευρωπαίους καταναλωτές να περάσουν προς μια πιο ισχυρή και πιο κυκλική οικονομία όπου οι πόροι χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο, αυξάνουμε την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση και αυτό έχει θετικές επιπτώσεις και για την οικονομία και στο περιβάλλον. Αυτή η έκθεση θέλει να προωθήσει αυτή η συζήτηση για το ρόλο της πολιτικής συνοχής στην, κατά την προώθηση και την εφαρμογή της κεντρικής ε, οικονομίας. Ε, μιλάμε ε, για 5,5 δισεκατομμύρια που δίνει η πολιτική συνοχή ε, για αυτό το θέμα, επομένως παίζει σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει όμως να αξιολογήσουμε το κατά πόσο χρησιμοποιούνται σωστά στα διάφορα κράτη-μέλη αυτά τα κονδύλια ε, και για να τα χρησιμοποιήσουμε αυτήν την αξιολόγηση στις διαπραγματεύσεις για την περίοδο μετά το 2020. Επίσης, ε, το Ταμείο Συνοχής ε, θα πρέπει να συνδυαστεί με το ορίζοντα 2020. Ε, μιλάμε για 550 εκατομμύρια για διάφορα project, καθώς και η οικονομία και οι επενδύσεις που κάνουν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο. Όλα αυτά. Στην έκθεση του συναδελφού προ... προτείνεται μία κυκλική, ολιστική θεώρηση της κυκλικής οικονομίας. Πέρα από την απλή διαχείριση των αποβλήτων και συμπεριλαμβάνει και τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι πράσινες ε, δημόσιες προμήθειες, η διαχείριση των λιμάτων, ε, βιοκαύσιμα, έρευνα, ανάπτυξη και κοινοτομία. Θεωρώ ότι μια πραγματική ενεργοποίηση των νομοθετικών μέτρων που προτείνει η Κομισιόν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και μια πραγματική ενημέρωση προς τους πολίτες για να γνωρίζουν πολύ καλύτερα τη σημασία των θεμάτων για τη δική του ζωή και για τις επόμενες γενιές. Αυτή η ενημέρωση είναι σημαντική και για τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Πριν από λίγους μήνες ε, έκανα ένα, υπέβαλε ένα ερώτημα προς τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζο της Κομισιόν για να δούμε αν το πλαίσιο για την, τις, ενισχύσεις, τις για το περιβάλλον, για την πουλια, απουλία για 60 εκατομμύρια ευρώ που είχαμε δώσει στην περιοχή αυτή της Ιταλίας για να περάσουμε ε, σε μια πιο κυκλική οικονομία. Ε, Μιλάμε τώρα για την επεξεργασία και τη διαχείριση των αποβλήτων. Η απάντηση τη Κομισιόν ήταν σαφή. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ενεργειακή αποδοτικότητα, λένε οι Βρυξέλλε, ε, αφορούν τομεί ε, τη οικονομία που σκοπό έχουν την προστασία του περιβάλλοντο, την ε, εξοικονόμηση τη ενέργεια, τη μείωση του διοξίδου του άνθρακα και σε παραγωγικού τομεί που δεν μολύνουν. Διαβάζω το κείμενο, λέξη-λέξη. Μιλάμε για παρεμβάσεις που σκοπό έχουν να αυξήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των ε, εργοστασίων, εγκαταστάσεων κτλ. Και, τα, και των υλικών. Ε, να ανακτώνται τα υλικά, να ανακυκλώνται τα υλικά και επομένως ε, εδώ δεν ε, συμπεριλαμβάνουμε την συλλογή και την διάθεση σε χωματερές των αποβλήτων. πρόκειται για σημαντική επιβεβαίωση της Κομισιόν. Η προστασία του περιβάλλοντος, η κυκλική οικονομία δεν έχουν καμία σχέση με τη χρηματοδότηση χωματερών και αποτεφρωτών. Επομένως, θα πρέπει να μην προωθούμε μέσω αυτής της έκθεσης ε, τρόπους ε, που μολύνουν το περιβάλλον. Ε, θα πρέπει να προωθούμε την ανακύκλωση των υλικών, την, ε, την επαναχρησιμοποίηση και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτά θα πρέπει να προωθεί η έκθεση. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ για τις ε, δηλώσεις των σκιωδών. Η κυρία Σπυράκη ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους, ε, τον γνωμοδότη, καθώς, τον εισηγητή, καθώς επίσης ε, και τους κυριαδείς για αυτό το έργο, το οποίο είναι ύψη τη σημασίας για τις Τοπικέ περιοχές, για τις περιφέρειες. Είναι σημαντικό όμως να παρουσιάσουμε διάφορες προτάσεις ε, κατά τόπους ε, με βάση ε, στη χρηματοδότηση που θα προέρχεται από το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα και επίσης είναι σημαντικό να καταλάβουμε ε, ότι υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα οικεία, όχι μόνο με την ε, κυκλική οικονομία ως ένα πλαίσιο, αλλά γενικότερα με την έννοια της κυκλικής οικονομίας. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να αναφέρω κάποια ζητήματα τα οποία θα ήθελα να συμπεριληφθούν στην έκθεση για την ε, κυκλική οικονομία, παρόλο που δεν υπάρχει μια ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Έχουν υπάρξει ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ε, οι οποίες υποστηρίζουν ε, έργα ε, για την κυκλική οικονομία, όπως είναι για παράδειγμα ο προϋπολογισμός 370 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος υποστηρίζει έργα καινοτομίας για την κυκλική οικονομία. Επίσης ε, χρηματοδοτούνται με 32 εκατομμύρια ε, ευρώ ε, και άλλα έργα για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει αναφορά στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία διότι δίνει παραδείγματα προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την κυκλική οικονομία. Επίσης θα ήθελα να υπάρξει αναφορά το έργο της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας για την κυκλική οικονομία όλα αυτά θα υποστηρίξουν ε, τους ιετέ, ε, θα υποστηρίξει ε, τις τοπικές αρχές για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν έργα κυκλικής οικονομίας. Βέβαια, αυτό δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τα ταμεία συνοχής και θα αποτελέσει μια σημαντική στρατηγική για όλους μας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν δοθεί 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να τονίσω ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε τις συγκεκριμένες ε, πρωτοβουλίες ε, και ε, τα ζητήματα τα οποία αφορούν την πολιτική μετά το 2020. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξουν τροπολογίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν το συγκεκριμένο Συμφωνώ λοιπόν ότι η στρατηγική ε, για τα πλαστικά είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι για την κυκλική οικονομία, διότι βρισκόμαστε ακόμα μονάχα στην αρχή και συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του κυρίου Γιακουβίτς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάουαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε η βιώσιμη οικονομία και η κυκλική οικονομία αναμφίβολα αποτελούν κομμάτι του μέλλοντος και το μέλλον είναι κάτι ε, το οποίο θα πρέπει να ε, χαρτογραφήσουμε. Ένα από τα πράγματα λοιπόν τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εδώ πέρα είναι ότι δεν αφορά μονάχα την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αλλά σε έναν βαθμό να θέσουμε ένα νέο πλαίσιο ε, και να εξετάσουμε τα συγκεκριμένα προγράμματα σχετικά με το αν είναι πράγματι κυκλικά και βιώσιμα έχω δει αρκετές προτάσεις ε, ε, για ε, προγράμματα τέτοιο, σαν αυτά. Όμως προγράμματα τα οποία εν τέλει αποδεικνύονται αρνητικά, είναι κατά της επαναχρησιμοποίησης και δεν ανοίγουν τον δρόμο προς την κυκλική οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν να τα ξέρουμε όλα αυτά όταν θέτουμε τα κριτήρια για να αξιολογήσουμε τα συγκεκριμένα προγράμματα. Και φυσικά η πραγματική δυσκολία που στοιχιώνει τις αγορές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης φαίνεται στη σελίδα 4. Μέχρι στιγμής υπάρχει ελλειπή ζήτηση ε, για υπηρεσίες κυκλικής οικονομίας διότι πολύ συχνά είναι πιο ακριβά από αυτά της γραμμικής οικονομίας ή τα ωφέλη δεν συνυπολογίζονται. Και φυσικά αυτή, αυτό είναι, ε, αυτή είναι η, απάτη. Πώς είναι δηλαδή δυνατόν να υποστηρίσουμε μια αγορά σε μετάβαση ε, από την γραμμική στην κυκλική οικονομία, πώς μπορούμε να στηρίξουμε την ζήτηση για κυκλικά προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα αυτά δεν είναι δωρεάν, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις δημόσιες συμβάσεις σε αυτόν τον ε, τομέα, θα απαιτήσουν μια αναγνώριση αυτών των αρνητικών στοιχείων ε, στα αγγλικά ε, θα έλεγα ότι αυτό είναι το ε, κοινωνικό κόστος της γραμμικής οικονομίας. Πώς λοιπόν θα πάρουμε αυτό το κόστος και θα το εφαρμόσουμε διότι το τίμημα, η τιμή για την πολιτική συνοχή είναι να διασφαλίσουμε ότι οι βιομηχανίες που αναπτύσσονται σε τομείς οι οποίοι θα πρέπει να αρθούν στο επίπεδο της υπόλοιπη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ε, γίνει αυτό στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομία και θα λειτουργήσει για τι περιοχέ αυτέ μονάχα σε περίπτωση που υπάρχει και μια αγορά για τα προϊόντα που παράγουν και γι' αυτόν τον λόγο αναφερόμαστε, αναφερόμαστε στα στοιχεία τη αγορά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την επιτυχία τη συγκεκριμένη ε, ε, περιοχή και γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ευθυγράμμιση με διάφορου τομεί τη Ευρωπαϊκή Πολιτική πέραν της συνοχής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο Βανίστερ Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια πράγματα τα οποία αναφέρθηκαν ήδη και πράγματι μιλήσαμε για την πολιτική συνοχή, αναφέρθηκε από πολλού. Όμως αν δεν εξετάσουμε την αγορά και ε, τα όσα μπορεί να ε, προσφέρει και να ζητήσει η αγορά, πριν ε, λίγο καιρό αναφέρθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει για νέα υλικά συσκευασιών που είναι πιο βιώσιμα και ότι όλο αυτό τώρα εισάγεται στην αγορά. Βλέπετε όμως ότι έχουμε, ε, έχει περάσει από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από πανεπιστήμια, έχει πλέον εισέλθει στην αγορά και η προώθηση η οποία απαιτείται για να καλύψουμε τις ε, συγκεκριμένες συσκευασίε για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ε, το καθιστούν πολύ πιο ακριβό. Από τις, από τις παλιές ε, πλαστικές συσκευασίε. Τι συμβαίνει λοιπόν. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει τα κεντρικά της στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει μισό λεπτό όλο αυτό θα είναι πολύ ακριβό. Δεν το κάνουμε λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει λοιπόν στη συνέχεια ένα πρόβλημα, διότι παράγουμε πολύ καλή νομοθεσία, η οποία στη συνέχεια όμως ε, δεν μπορεί να ε, αποφέρει αποτελέσματα. με αυτήν την νέα περίοδο θα πηγαίναμε στην ε, κυκλική οικονομία όπως υπόθηκε όμως ε, θα πρέπει εάν ε, φέρουμε τα πράγματα πολύ γρήγορα θα έχουμε προβλήματα. Πρώτα πρέπει να σκεφτούμε καλά. Επίσης τα βιοδιασπόμενα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορα πράγματα. Παίζεις με κάτι στην παραλία το οποίο τελικά καταλήγει στην θάλασσα και καταλήγει σε αυτά τα νησιά πλαστικής σούπας σε όλο τον κόσμο. Ε, τι ε, κανόνες λοιπόν εφαρμόζονται εδώ πέρα. Τίποτα απολύτως, ε, καμία βάση λοιπόν δεν υπάρχει για να εγκριθούν τα συγκεκριμένα διασπόμενα υλικά. Μπορεί να έχουμε ένα φυτό το οποίο, το οποίο φυτεύουμε και στη συνέχεια η ίδια η γλάστρα διαλύεται από το ίδιο φυτό. Όμως δεν το κάνουμε διότι κοστίζει 2 σεντ παραπάνω. Τι κάνουμε λοιπόν, δημιουργούμε διάφορες νομοθεσίες νομοθεσίες ε, χωρίς να τις ακολουθούμε και χωρίς να μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και αυτό δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Ε, Κοιτάζοντα την εισαγωγή στην αγορά, σκεφτόμαστε ότι η αγορά θα τα λύσει όλα και βλέπουμε όμω τελικά ότι η αγορά δεν το κάνει διότι είναι πολύ ακριβό, είναι πιο ακριβό. Ε, μπορούμε λοιπόν να βγάζουμε εδώ πέρα νομοθεσίας. Ε, είμαι υπέρ της εξάντε διαδικασίας, όμως θα πρέπει να τονίσουμε ε, ότι ε, να τονίσουμε στην Κομισιόν ότι ε, οι περιοχές, οι περιφέρειες θέλουν να το κάνουν αυτό, αλλά στο σκεφτούμε λιγάκι καλύτερα. Ας βρούμε κάποιες τροπολογίες λοιπόν, διότι είναι σημαντικό όλο αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει λιγάκι να επιβραδύνουμε. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση του κυρίου Σκέρλετς είναι πολύ σημαντική και τα μήνυματά της επίσης ε, πολύ αξιόλογα και σημαντικά. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια στάση και να σκεφτούμε αν θα πρέπει να συνεχίσουμε τη μέχρι τώρα πολιτική ή να την αλλάξουμε. Και δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Αυτό είναι αυτονόητο μπορούμε να έχουμε να χρησιμοποιούμε ξανά οτιδήποτε. Το θέμα είναι να μην πετάμε κάτι που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και αυτό θα πρέπει να, να χτίσει υποχρέωση. Αλλά αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη από τη φάση του σχεδιασμού και της παραγωγής. Θα πρέπει ήδη στην φάση του σχεδιασμού να προβλέπουμε τη μεταγενέστερη χρήση του προϊόντος και την επαναχρησιμοποίησή του. Επίσης, ό,τι αφορά την, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Για παράδειγμα, θα πρέπει να επεκτείνουμε τη χρήση της ηλιακής ενέργειας ή να αναζητήσουμε άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μήπως θα πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο την πυρηνική ενέργεια και να περιορίσουμε τις επενδύσεις στην αιωλική και την ηλιακή ενέργεια, για παράδειγμα. Εδώ νιώθω μια πολιτική του Κάτσα και καρτέρα, wait and see. Ε, για δέκα χρόνια δούλευα σε μια εταιρεία που παρήγε ε, αντλίες ε, για νέα χρήση διζελοκινητήρων. Υπάρχει αυτή η παράδοση λοιπόν και υπάρχουν τεχνολογίες για επαναχρησιμοποίηση τέτοιων κινητήρων για παράδειγμα ή συστοιχειών ε, μπορούμε μπαταρίες που έχουμε χρησιμοποιήσει να προβλέψουμε να επαναχρησιμοποιούνται. Πιστεύω ότι και αυτό το θέμα θα μπορούσε να το λάβει υπόψη η έκθεση. Τη σήμερα ημέρα βέβαια οι εταιρείε δεν ενδιαφέρονται πολύ για επαναχρησιμοποίηση ούτε η αυτοκινητοβιομηχανία ούτε άλλη παραγωγή προϊόντων. Γιατί όσο περισσότερο χρησιμοποιείται μια μηχανή, ένας κινητήρας, ε, ε, τόσο λιγότερο κερδίζει ο παραγωγός. Ε, είχαμε την περίπτωση των αυτοκινήτων Volvo, ακριβώς επειδή είχαν μακριά ζωή και μπορούσαν να κυκλοφορούν και να χρησιμοποιούνται χωρίς πρόβλημα για πολλά χρόνια. Φυσικά η Volvo δεν ε, αποκόμισε τα αναμενόμενα κέρδη. Και γι' αυτό είναι κάπως επιφυλακτική η παραγωγή για τη μακρά χρήση ζωής των προϊόντων τους. Θα πρέπει όμως να καταπολεμήσουμε την απόρριψη των προϊόντων με την πρώτη ευκαιρία και μόνο επειδή ένα ανταλλακτικό τους έχει καταστραφεί. Έχουμε πραγματικά πεδίο δόξης λαμπρό με την ε, κυκλική οικονομία και θα μπορούσαμε να περιορίσουμε αυτή την αμυγός οικονομική προσέγγιση στα πράγματα, να εθετήσουμε μια πιο σφαιρική προσέγγιση. Αλλιώς θα καλούμαστε να αλλάζουμε κάθε χρόνο τις οικιακές μας συσκευές ή τα αυτοκίνητά μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποια λογικά όρια και προδιαγραφές και πρότυπα. γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε και τη φορολογική πολιτική μας, δίνοντας κίνητρα φορολογικά. Για να σταματήσουμε να ενισχύουμε την αγορά νέων προϊόντων, αλλά να επαναχρησιμοποιούμε τα παλιά περισσότερο. Κύριε Μπρέσο, ευχαριστώ. Δεν θέλω να πάρω τον λόγο, γιατί έχουμε να μας εκπροσωπεί η σκιώδηση συγγήτρια μας. Ε, αλλά εγώ έχω ασχοληθεί προσωπικά επί 30 χρόνια με την κυκλική οικονομία και συμμετείχα και στην ομάδα υψηλού επίπεδου που εργάστηκε για να προετοιμάσει τα έγγραφα για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Από τη θέση βέβαια του μέλους της ε, Επιτροπής των Περιφερειών, όχι ως Ευρωβουλευτής. Θα ήθελα λοιπόν με αυτή την ιδιότητα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες θεωρώ ότι είναι εκ των ονουκάνευ. Να επενθυμίσουμε ότι όταν μιλάμε για την κυκλική οικονομία, μιλάμε για μια τάση την οποία δεν θα πετύχουμε ποτέ, γιατί υπάρχει η, η εντροπία της α, ενέργειας και της ύλη. Μιλάμε για τα διάφορα βήματα τα οποία λείπουν και τα οποία μας αποτρέπουν, δεν μας εμποδίζουν να φτάσουμε στην πλήρη κύκλικη οικονομία. Είναι μια τάση λοιπόν. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που λένε ότι οι μηχανισμοί που μπορούν να μας επιτρέψουν να επιταχύνουμε την διαδικασία είναι κυρίως οι μηχανισμοί των κινήτρων που βασίζονται σε κίνητρα. Οι κανόνες βοηθάνε, εξυπηρετούν, αλλά κυρίως βοηθάνε τα κίνητρα, το να δώσουμε κίνητρα. Γιατί μας οθούν προς το σχεδιασμό προϊόντων και κυρίως συσκευασιών που μπορούμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε εύκολα, να τα ανακυκλώσουμε εύκολα και πρακτικός πώς αλλά και οικονομικός πώς. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μια πράσινη λογική, ένας πράσινος σχεδιασμός των προϊόντων. Και κοιτάξτε, δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν θετικές τάσεις και αρνητικές τάσεις. Φερρυπίν. Στον τομέα της, ε, των αυτοκινη, της αυτοκινητοβιομηχανίας όλο και μεγαλώνουν τα αυτοκίνητα. Έχουμε όλο και πιο περίπλοκα υλικά ενσωματωμένα στα αυτοκίνητα. Και με αυτόν τον τρόπο είναι αδύνατο να τα επισκευάσουμε, να τα επιδιορθώσουμε τα αυτοκίνητα τα προϊό... και πολλά άλλα προϊόντα. Είναι τόσο περίπλοκα, τόσο σύνθετα, με σπάνιες πρωτεσίλες, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα επισκευάσουμε. Να επισκευάσουμε και τα ανταλλακτικά τους, ας πούμε. Επομένως δεν είναι αλήθεια ότι κινούμαστε σαφώς προς την κυκλική οικονομία. Δεν ισχύει αυτό. Πέρα από τους υποχρεωτικούς κανόνες, πάνω απ' όλα ε, αυτό που είναι σημαντικό είναι τα κίνητρα, ειδικά για τις συσκευασίε. Μέχρι στιγμής οι χρήστες των πρώτων δευτερογενών υλών, που προέρχονται δηλαδή από την ανακύκλωση των προϊόντων, οι πρώτοι που το κάνανε ήταν οι Κινέζοι. Και μέχρι που αρχίσαν να έχουν δικά τους πρωτογενή, ε, πρώτες μάλλον δευτερογενείς ύλες. Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Απλώς εξάγουμε υλικό προς ανακύκλωση. Δεν είμαστε καν σε θέση να το κάνουμε εσωτερικά, να κάνουμε λέει, την ανακύκλωση του εσωτερικού της Ευρώπης. Επομένως πρέπει να δώσουμε ε, κίνητρα, παροχές, ε, για να υπάρξουν εταιρείε που προωθούν αυτή την ανακύκλωση. Γιατί αλλιώς δεν τα καταφέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε. Επομένως, εγώ δεν είμαι και τόσο αισιόδοξη, γιατί έχουμε θετικά φυσικά στοιχεία και μηνύματα, αλλά υπάρχουν και πολύ αρνητικά. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγάλη έμφαση στα κίνητρα παρά στις περίπλοκες νομοθεσίες, δεσμευτικές κτλ, οι οποίες τελικά δεν γίνονται σεβαστέ και δεν εφαρμόζονται από κανέναν. Αλλά όπως σας είπα, δεν είμαι και τόσο πεπισμένη ότι κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση. Γιατί τα περισσότερα σημερινά προϊόντα είναι πάρα πολύ περίπλοκα, πάρα πολύ σύνθετα ως προς τη σύνθεσή τους και για να τα διαλύσουμε ας πούμε και να μπορέσουμε να ανακυκλώσουμε κάποια ανταλλακτικά ας πούμε, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο να κυκλώσει κανείς ένα αυτοκίνητο που έχει, δεν ξέρω εγώ πόσα, τα περισσότερα εξαρτήματά του ηλεκτρονικά. Είναι πολύ πιο εύκολο αν είναι μηχανικό το αυτοκίνητο. Γιατί όταν είναι εύκολο μπορεί να αντικαταστήσει ένα κομμάτι ας πούμε, του όλου, του αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε προϊόντο. Ενώ όταν είναι πολύ σύνθετο τελικά το πετά και αγοράζει άλλο. Είναι πολύ σύνθετο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να έχουμε κανόνες και νομοθεσία, αλλά αν δεν έχουμε κίνητρα, δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχουμε αποτελέσματα. Ε, απλώς κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι κάτι πετυχαίνουμε. ζητώ συγγνώμη που τα λέω αυτά, ήθελα να πω στον εισηγητή μας να το, να το σκεφτεί αυτό το, πράγμα και να δώσει σημασία στα κίνητρα ε, και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Αυτά ήταν τα σχόλια των μελών της Επιτροπής Ρέτζι και τώρα θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Νεοντίνοβα. Καταρχάς, θα ήθελα ε, και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ ε, τον εισηγητή για την έκθεσή του. Πραγματικά πιστεύουμε ε, ότι είναι ένα πολύ καλό κείμενο το οποίο αντικατοπτρίζει την μεγάλη σημασία της κυκλικής οικονομίας για τις περιφέρειες και όπως βλέπουμε προκάλεσε μια έντονη συζήτηση το οποίο επίσης είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Ε, προφανώς η πολιτική ε, συνοχή ε, συνεισφέρει έντονα στην κυκλική οικονομία ε, και όπως έχει αναφερθεί ορθά ε, η ε, κυκλική οικονομία δεν προβλέπεται στους κανονισμούς όμως η ιδέα της κυκλικής οικονομίας υπάρχει εκεί πέρα έχουμε μια αποτελεσματικότητα πόρων και επίσης η σκέψη, η ιδέα της κυκλικής οικονομίας αλλά και η εφαρμογή αυτής ή βρίσκονται ε, ήδη ε, στα ε, λειτουργικά μας προγράμματα. Αυτό όσον αφορά τα απορρίμματα, αλλά και χάρη στην εκ των προτέρων ερεσιμότητα υποστηρίζουμε περισσότερες παρεμβάσεις στον στην ιεραρχία των αποβλήτων, δηλαδή περισσότερη ανακύκλωση. Επίσης ε, έχουμε την ε, συγκεκριμενοποίηση των αποβλήτων και αυτό επίσης είναι ένας ε, τρόπος για, τρόπος για να προωθήσουν οι περιφέρειες από κάτω προς τα πάνω την έρευνα που πρέπει να γίνει. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όχι μονάχα για την καινοτομία στην περιοχή αλλά ταυτόχρονα και για την ε, διαπεριφερειακή συνεργασία και ειδίκευση. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με ε, περιφέρειες σε διάφορες, ε, σε διάφορους τομείς διότι ε, η συνεργασία αυτή, ε, αν ασχοληθούμε με αυτό μονάχα σε μια περιφέρεια, δεν θα επέλθει ε, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο χρειαζόμαστε. Εργαζόμαστε λοιπόν για να ενώσουμε, τις, να συνδυάσουμε τις περιφέρειες με τις διάφορες προτεραιότητες. Αυτό βρίσκεται λοιπόν στο επίκεντρο της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας που είναι ήδη διαθέσιμη. Επίσης, η κυκλική οικονομία δεν αφορά μονάχα τα απορρίμματα και η κοινοτομία, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις ανανεώσιμες. Επίσης, αφορά σε μεγάλο βαθμό το ε, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την ενίσχυση αυτών ε, για να για την εξέβρεση λύσεων και χάρηκα ιδιαιτέρως ε, που άκουσα την αναφορά ε, σχετικά ε, με τις καινοτομίες που υπάρχουν. Έχουμε όντως πάρα πολλές καλές καινοτομίες που υποστηρίζουμε μεταξύ αυτών η κυκλική οικονομία. Επίσης θα ήθελα να χαιρετήσω το έργο το οποίο γίνεται για, την, αγροτική, για το αγροτικό θεματολόγιο. Εκεί υπάρχουν κάποιες συνεργασίες και και στον τομέα της κυκλικής οικονομίας όπου διάφορες πόλεις συνεργάζονται για τις προκλήσεις που εμφανίζονται ε, και μία από αυτές τις εταιρικέ ε, σχέσεις αφορά και την κυκλική οικονομία. Έχουμε επίσης την ποιότητα αέρα. Ε, αυτά λοιπόν όλα έρχονται και προστίθενται στα έργα τα οποία αναφέρθηκαν σήμερα. Φυσικά υπάρχουν πολλά ωφέλη και πλεονεκτήματα, δεν τελειώνουμε όμως εκεί. Πολλά ακόμα έχουν ε, να γίνουν. Ε, λυπάμαι όμως ε, για το γεγονό ότι υπάρχει έντονη έμφαση ε, για το γεγονό ότι δεν είναι δυνατόν το παρόν νομοθετικό πλαίσιο να συμπεριλάβει την πραγματική συνεισφορά τη κυκλικής οικονομίας. Έχει αναφερθεί και αυτό στην έκθεση, συγκεκριμένα στη σελίδα 9 ε, ε, καταλαβαίνω ότι ε, θέλουμε να υπολογίσουμε, να μετρήσουμε ακριβώς το πλαίσιο της παρέμβασης. Ναι βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ακριβή συνεισφορά της πολιτικής συνοχής, όμως είναι πολύ δύσκολο να έχουμε επακριβή στοιχεία, διότι θα είναι δύσκολο να υπολογίσουμε την τη συνεισφορά μας. Το πιο σημαντικό αφορά την εφαρμογή και τι συμβαίνει κατά τόπους Πιστεύω λοιπόν ότι ε, η κριτική είναι ορθή, όμως ε, δεν θα πρέπει να τονίζεται σε τέτοιο ε, βαθμό, διότι πιο σημαντικό είναι το τι συμβαίνει κατά τόπους παρά το πώς μετρώνται τα πράγματα και τώρα για την περίοδο μετά το 2020 κάποια πράγματα ναι μπορούν να βελτιωθούν. Θα δείτε την πρότασή μας τον Μάιο, όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι η κυκλική, η κυκλική οικονομία ε, είναι μια μετάβαση, ε, μια μεταμόρφωση των οικονομιών μας που πρέπει να λάβει χώρα και δεν θα είναι κάτι εύκολο. Ε, είναι αληθές ότι απαιτείται ένα συνδυασμός νομοθετικών εργαλείων και επίσης είναι αληθές ότι ε, η ε, δημόσια παρέμβαση όσον αφορά την χρηματοδότηση θα είναι αναγκαία, όπως είναι για παράδειγμα η πολιτική συνοχή, όμως ε, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι ναι έχουμε μεγάλη συνεισφορά πάνω σε αυτό, δεν είναι εύκολο είναι ε, μια ε, μεγάλη πρόκληση του συγκεκριμένου όργα, έργο όμως είναι και σημαντικό για την ε, μετάβαση μετά το 2020 που πρέπει να λάβει χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Σιγητά, κύριε Σκύρλετς, θέλετε το λόγο για να δευτερολογήσετε μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Παρακαλώ. Ο κύριος Σκύρλετς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ λακωνικός να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις πολύ εύστοχες προτάσεις τους και πολύ χρήσιμες. Ε, επί του παρόντος το πρόβλημα έγκυται στο ότι με βάση τις στατιστικές και τις διατάξεις δεν έχουμε κοινό ορισμό για, το, για την κυκλική οικονομία και έτσι δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε τη συμβολή της θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να συγκεντρωθούν ε, κατάλληλες πληροφορίες και για να προσελκύσουμε τις επενδύσεις βέβαια, αλλά όχι μόνο για την ε, αξιοποίηση, εκμετάλλευση των αποβλήτων, ε, αλλά και για άλλα μέτρα. Και θα πρέπει να επεκταθούμε και σε άλλους τομείς που μπορούν να καλύπτονται από την έννοια της κυκλικής οικονομίας. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς με διάφορα κίνητρα, με ενάυσματα, ίσως με φορολογικά κίνητρα ή πώς, ίσως με κάποια φορολογική μεταρρυθμίση να δώσουμε τα ενάυσματα, ώστε να γίνει μια μετάβαση, μια αλλαγή της αγοράς και οι καταναλωτές όλο και περισσότερο να προσανατολίζονται σε προϊόντα που προέρχονται από δευτερογενείς πρώτες ύλες. και αυτό εντάσσεται σε κάποια καλά στοιχεία της διαχείρισης ή διάθεσης αποβλήτων. Να δημιουργήσουν δηλαδή δευτερογενή, ε, δευτερογενείς πρώτες ύλες. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε την πολιτική μας προκειμένου να προωθήσουμε νέο τρόπο σκέψης για την παραγωγή προϊόντων, ώστε να έχουν μακρύτερη διάρκεια ζωής, να, ε, αλλά να μπορούμε να τα αλλάξουμε ελεύθερη, να τα επαναχρησιμοποιήσουμε και αν πραγματικά φτάνουν στο τέλος της ζωής τους και δεν μπορούν πια να χρησιμοποιηθούν, να μπορούμε να ε, προσανατολιστούμε σε άλλα ή να μπορούμε να αλλάζουμε μόνο κάποια ανταλλακτικά τους ε, για να μην τα καταργούμε πλήρως. Ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση, επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα και σημαντικός άξονας της κυκλικής οικονομίας ε, η ενεργειακή απόδοση. Επίσης η βιοοικονομία και φυσικά ο περιορισμός των πλαστικών, σήμερα ο όγκος τους είναι ακόμη τεράστιος, αλλά καλό θα ήταν να κάνουμε ένα βήμα πρόοδου και να αλλάξουμε ε, ε, την οικονομία μας και να περάσουμε από τα ορυκτά καύσιμα σε δύο καύσιμα και να αναπτύξουμε και νέα υλικά που θα έχουν παρόμοια ή ακόμη και καλύτερη χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν τα μέχρι τώρα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση αυτή, ε, την εξέταση του σχεδίου Προτείνω διορία για την κατάθεση τροπολογιών μέχρι στις 11 Απριλίου 12 το μεσημέρι. Τετάρτη 11 Απριλίου 12 το μεσημέρι λίγη η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Και ολοκληρώσαμε τη συζήτηση της εκθέσεως ε, Σκέλετς και θα περάσουμε στην επόμενη συζήτηση στο σημείο 5 που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων επί της εκθέσεως πρωτοβουλίας με θέμα την πρόθεση της οικονομικής ανάπτυξης και της συνοχής της παραμεθόριας περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρυσι τον Οκτώβριο η Επιτροπή υιοθέτησε μία μη νομοθετική ανακοίνωση με θέμα την πρόθεση της οικονομικής ανάπτυξης και της συνοχής στις ευρωπαϊκές παραμεθόριες περιφέρειες. Οι παραμεθόριε περιοχέ έχουν λιγότερη οικονομική ανάπτυξη από τι υπόλοιπε Η ανακοίνωση τη επιτροπή εστιάζεται σε 10 σημεία στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μπορούν να περιορίσουν την περιπλοκότητα, το μήκο και το κόστο των διαμεσοριακών συναλλαγών και να προωθήσουν τη συγκέντρωση υπηρεσιών εντό των εσωτερικών σύνορων. Η Επιτροπή μα αποφάσισε να συντάξει έκθεση πρωτοβουλία πέρυσι το Δεκέμβριο. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από την Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών το Μάρτιο και περιμένουμε την έγκριση της ε, Διάσκεψης Προέδρων, ε, των Προέδρων τον Απρίλιο. Δύο επιτροπές αποφάσισαν να εκπονήσουν έκθεση. Οι επιτροπές απασχόλησης και ε, πολιτισμού, θα, συγγνώμη, θα γνωμοδοτήσεις, ενώ ε, εμείς αναθέσαμε την έκθεση πρωτοβουλία στον κύριο Ξίστοφ Χέτμαν από το ΕΛΚ, που θα μας κάνει την πρωταρχική παρουσίαση σήμερα και θα μας υποβάλει, αν δεν κάνω λάθος, το σχέδιο έκθεσή του το Μάιο. Έχω δίκιο, μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Χέτμαν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα αυτό των παραμεθόριων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα που επιδέχεται μακροσκελού συζήτηση εκτενέστατης δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα θέμα. Θα μπορούσε να επεκταθεί σε περισσότερα θέματα και σε περισσότερε μέρε συζήτηση. Πάντω είναι σημαντικό να τονίσουμε και την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την δική μα προσπάθεια στα πλαίσια τη έκθεση πρωτοβουλία που πραγματικά υπογραμμίζουν, επισημαίνουν αυτή την κατάσταση, διαπιστώνοντα ότι οι παραμεθόρειε περιφέρειες ακριβώ εξαιτία τη θέση του, αντιμετωπίζουν κάποιες ε, ιδιαίτερες προκλήσεις. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποδώσει δέωσα προσοχή και να δώσει ξεχωριστή υποστήριξη σε αυτές τις παραμεθόριες περιφέρειες. Βέβαια δεν υπάρχει ένα καλούπι για τις παραμεθόριες περιφέρειες, δεν υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά υπάρχουν ιδιαιτερότητε και οι λύσει θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτέ τι ιδιαιτερότητε. Έχουμε κάποιε παραβεθόρε περιοχέ ε, στι οποίε ε, ε, επικρατούν καλέ συνθήκε, ενώ άλλε που είναι πολύ περιφερειακέ και απόκεντρε αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και αντιμετωπίζουν και ένα πραγματικά οξύ δημογραφικό πρόβλημα. Α μην ξεχνούμε ότι οι παραμεθόριες περιοχές καταλαμβάνουν περίπου το 40% της ευρωπαϊκής επικράτειας. Επίσης έχουν πληθυσμό γύρω στα 150 εκατομμύρια κατοίκου. Δηλαδή είναι το 30% του, επίσης του ΑΕΠ, του κοινοτικού ΑΕΠ. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υπάρχει η σημαντική πρόταση ότι ακόμη και αν, αν καταργούσαμε όλα τα εμπόδια σε σχέση των, περιφε... παραμεθόριων αυτών, ε, οι περιφέρειες αυτές θα αύξαναν κατά 8% τον πλούτο τους, το ε, ακαθάριστο προϊόν, το τους. Ακόμη και η μείωση κατά 20% των ε, ε, εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες αυτές, το ΑΕΠ τους θα, αυξανόταν κατά 2%. Βλέπετε ότι και με μια μικρή πρόοδο μπορούμε να βοηθήσουμε τις περιφέρειες αυτές. Το 1990 η πρωτοβουλία Interreg της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας στις παραμεθόριες περιφέρειες αφιέρωσε 6 ε, δισεκατομμύρια ευρώ στο θέμα αυτό και θα πρέπει να επενέσουμε αυτό το πρόγραμμα γιατί λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες ε, των παραμεθόριων περιοχών. Στην δική της ανακοινώση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει τους σημαντικότερους τομείς που χρήζουν επεξεργασίες και που ταλανίζουν τις ε, περιοχέ, περιοχές. Για παράδειγμα, εντατικοποίηση της συνεργασίας, τελειοποίηση της νομοθετικής διαδικασίας, δυνατότητα διασυνοριακής ε, δημόσιας διοίκησης, διευκόλυνσης της διασυνοριακής πρόσβασης και προώθηση της καλύτερης συμπληρωματικότητας στις ε, υπηρεσίες υγείας. Εγώ θα πρόσθετα σε αυτά τα θέματα την ε, ε, ανάληψη οικονομικών δραστηριοτήτων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην οικονομική δραστηριότητα στις παραμεθόρειες αυτές και θα πρόσθεται επίση και το δημογραφικό ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή τη προτείνει αρκετέ ενδιαφέρουσε λύσεις για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των παραμεθόριων περιοχών. Για παράδειγμα, η δημιουργία, η δημιουργία ενιαίας πύλης ε, ε, για τις παραμεθόριες και οι χάρτες για την ε, διαπεριφερειακή συνεργασία, διασυνοριακή συνεργασία, διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας και κάποια πιλωτικά προγράμματα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και απαραίτητα. Πάντως, ε, οι παραμεθόρεις ε, περιοχές, παρά τις πρωτοβουλίες αυτές, εξακολουθούν να έχουν προβλήματα, εξακολουθούν να είναι σε μη προνομιακή θέση και αναπτύσσονται με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν μπορούμε πάντα να βρίσκουμε τις σωστές λύσεις για τα προβλήματά τους. Πάντως χαίρομαι για μία από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα επευκαιρία ευκαιρία της παρουσίας των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις για μερικά θέματα που πραγματεύεται η ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση προτείνονται κάποια βήματα για να εντοπιστούν ε, τα αποτελέσματα ε, που έχουν η χρήση των διαφόρων πρωτοβουλειών και μεθόδων. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η αποτίμηση. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα υποβάλει τα αποτελέσματα πιλωτικών προγραμμάτων ε, με αποδέκτες τους ε, δημόσιους φορείς, ώστε να, να επιληθούν κάποια νομικά ή διοικητικά προβλήματα που ταλανίζουν κυρίως τις διαμεθοριακές περιοχές. Σε τι φάση βρισκόμαστε ως προς αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης, ε, είπατε ότι θα γίνουν κάποιες μελέτες για, την, για τις σιδηροδρομικές διασυνδέσεις ε, έγιναν αυτές οι μελέτες για την ε, διασύνδεση και πότε θα περιμένουμε τα αποτελέσματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, ε, σε ό,τι αφορά την εδαφική συνεργασία για τη σχετική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόκειται για μία πρόταση που θα ήταν υποτίθεται το αντίδοτο όλων των προβλημάτων των παραμεθόριων περιοχών και μάλιστα αναφέρεται και στην τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι γίνεται με τις εργασίες αυτής της ε, ομάδας εδαφικής συνεργασίας. Επίσης, ε, σίγουρα μέχρι στιγμής έχουν αρθεί πολλά εμπόδια και έχει σημειωθεί πρόοδος. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν με αργούς ρυθμούς οι επενδύσεις και έχουμε μεν αρκετές καλές πρακτικές σε πολλές περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές περιοχές, αλλά όλα αυτά ένα μεγάλο τμήμα των παραμεθόριων περιοχών είναι περιφερειακές και εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται περιφερειακές περιοχές. Και σίγουρα έχουν πραγματοποιήσει πρόοδο, αλλά οι πιο ευμερούσες ε, περιοχές που δεν έχουν τέτοια προβλήματα μεθοριακά έχουν ακόμη σημαντικότερη ανάπτυξη. Επίσης, το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά το αλλά πιστεύω ότι χρήζουν μεγαλύτερη προσοχή και ενδιαφέροντο οι περιοχέ αυτέ και από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και από τα κράτη-μέλη και από τι ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης. Επίσης, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δείξουν μεγαλύτερη τόλμη και θάρρος. Και τέτοιες πληροφορίες δεν τις βρίσκουμε στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως θα είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν τέτοιου είδου πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να λύσουμε τα ιδιαίτερα, τα ιδιαίτερα προβλήματα των παραμεθόριων περιοχών. Γι' αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Πολύ συχνά κάποια κοινά διασυνοριακά προγράμματα και το δίκαιο, το ενωσιακό, εμ, ακριβώς εκλαμβάνεται ως απειλή στην εθνική κυριαρχία σε πολλές χώρες μέλη. Όπω είπα, η ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν περιλαμβάνει μια ανάλυση και αυτού του προβλήματο που κατά τη γνώμη μου είναι ένα ε, ουσιαστικό και απτό πρόβλημα που καλό θα ήταν να συζητηθεί. Αντίθετα, πιστεύω ότι αν δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ε, για την ανάληψη της ευθύνης από τοπικές και περιφερειακές αρχές, τότε θα μπορέσουμε να άρουμε πολλά εμπόδια που ακόμη υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι μία λέξη κλειδί που είναι απαραίτητη σε όλες τις δραστηριότητε της Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σμόλκοβα θα μας παρουσιάσει τη θέση του σκιώδου συγγετού. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Υποστηρίζουμε την ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση με τον ίδιο τίτλο. Οι μεθορικές περιοχέ είναι το 40% τη Ευρωπαϊκή Ένωση και 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εκεί. 30% ε, του ΑΕΠ ε, παράγεται σε αυτέ τι παραμεθόριες περιοχέ. <clears throat> και έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια καθημερινού επιβάτε που ταξιδεύουν μπρο πίσω κάθε μέρα, α πούμε. <clears throat> περιφερειακές μας, οι μεθοριακές μας περιοχές θα πάνε λιγότερο καλά γενικά από τις υπόλοιπες περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι δημόσιες υπηρεσίες, ε, σχολεία, νοσοκομεία είναι σε χειρότερη κατάσταση. Ε, αυτό είναι τεράστιο θέμα ε, για πολλούς πολίτες καθημερινά και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους. Οι πολίτες που ζουν στις μεθοριακές περιοχές θα μπορούν να είναι σε θέση να υποφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες ε, που προσφέρονται και από τι δύο μεριές των συνόρων. Συμφωνώ ότι δεν μπορούν να επιληφθούν όλα αυτά τα προβλήματα μόνο με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά έχουμε πετύχει πάρα πολλά μέσα από τα ταμεία και το πρόγραμμα Interreg. Ε, για αυτό λοιπόν, ε, αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν. Ε, παράλληλα, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συγχρονιστούν κάπως, ειδικά τα όμορα και να αντιμετωπίσουν ε, τα διοικητικά εμπόδια και, τις, ε, και τα νομικά κολλήματα που εμποδίζουν την καλή συνεργασία. Είναι επίκαιρη η παρέμβαση αυτού του Κοινοβουλίου, χαίρομαι που θα παρέμβουμε και περιμένω, προσβλέπω ε, σε μια πολύ εποφελή συνεργασία. Αυτά από το συνάδελφο που εκπροσωπώ, τον αντιπρόεδρο δηλαδή. Από το ECR δεν βλέπω κανένα Είμαι και εγώ σκιώδης εισηγήτρια και θα μιλήσω κι εγώ ε, στα βουλγαρικά, στη γλώσσα μου. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Είμαι η σκιώδης εισηγήτρια, όπως σας είπα, και ως τέτοια θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη δημόσια διαβούλευση που έγινε online για την προσέγγιση των μεθοριακών περιοχών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταγράψουμε όλα τα, τα εμπόδια που ταλανίζουν αυτές τις περιοχές. Η διασυνοριακή συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με το περιβάλλον, την απασχόληση, την κινητικότητα επίσης των εργαζομένων. Όμως κάποια στοιχεία αυτής της συνεργασίας δεν ε, υπάρχουν, εξού και η δύσκολη συνεργασία. Ως και ως εισηγήτρια λοιπόν του Άλντε θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτή την έκθεση, ε, μάλλον πάνω στην, σε μια έκθεση πρωτοβουλίας του 2016. Ε, χαίρομαι που οι συστάσεις που είχαμε εκδώσει τότε λύθησαν υπόψη τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ λοιπόν ότι η επιλογή της νομοθετικής πράξης ε, ως σωστή, τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τις συνθήκες αυτής της συνεργασίας ανάλογα με τις ανάγκες τους. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι οι προτάσεις να δημιουργηθεί μια, ένα τμήμα στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και η πλατφόρμα online είναι πολύ θετικά μέτρα. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει καλύτερο συντονισμός ε, για να καλυφθεί αυτή, αυτό το διοικητικό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο περιοχές των ε, συνόρων. Επίσης, η ηλεκτρονική διαχείριση θα διευκολύνει την διοικητική αυτή μεθοριακή συνεργασία. Σε ό,τι αφορά τα κενά, σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία, θεωρώ ότι η Eurostat και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να βελτιώσουν τη συνεργασία τους, ούτω ώστε να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Το Interreg παίζει σημαντικό ρόλο, καθοριστικό ρόλο και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω προσπάθειες για να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη όλων των μεθοριακών περιοχών. Αναμειγνύοντας σωστά τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης, είτε ευρωπαϊκής είτε εθνικής. Χαιρετίζω το ρόλο των εδαφικών αυτών ομάδων ανάπτυξης για την υποστήριξή τους και για το ρόλο που παίζουν ως πλατφόρμες για την ε, υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές μπορούν και αυτές να βοηθήσουν αυτές τις μακροπεριφέρειες να αντιμετωπίσουν ε, τα προβλήματα και τις προκλήσεις. Μπορεί να χρησιμεύσουν πάρα πολύ στις ε, μεθοριακές ε, περιοχές. Πολλές περιοχές έχουν τεράστια προβλήματα λόγω μετανάστευσης. Εξού και η ανάγκη να ενισχύσουμε την ανταλλαγή καλών πρακτικών για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτά ευχαριστώ. Και τώρα συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους σκιώδους εισηγητές. Η κυρία Άντερσον. Θα πάρει κάποιο το λόγο να την αντικαταστήσει. Όχι. Κύριε Νταμάτο τότε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάγκη να αυξήσουμε την, την ανάπτυξη αυτών των ε, μεθοριακών περιοχών. Και χαίρομαι για τη μέθοδο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μια διαβούλευση δημόσια που έγινε online σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έγιναν έρευνες και ανταλλαγές απόψεων με, τις, με τους ενδιαφερόμενους. Η Κομισιόν ε, έθεσε διάφορα ερωτήματα και προβληματικές ε, με βάση τις ανάγκες και τα προβλήματα που ζουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών και οι επιχειρήσεις. Ε, παρότι αυτά τα προβλήματα δεν αφορούν αποκλειστικά τις μεθοριακές περιοχές, αλλά παρόλα αυτά αυτές τα αισθάνονται πολύ περισσότερο, λόγω της συχνότητας και του επίπεδου αλληλεπίδραση αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε, μεταξύ τους δηλαδή. Η ανακοίνωση αυτή δείχνει ορισμένε περιπτώσεις για κάποια πρακτικά προβλήματα. Παραδείγματο χάρη την υγειονομική περίθαλψη ή το πρόβλημα των επαγγελματικών προσόντων, που σίγουρα θα πρέπει να, τα, ε, να εγγύψουμε από αυτόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, Περιμένω το σχέδιο έκθεση του συναδέλφου, αλλά προ το παρόν θα πρέπει να, να σα πω ότι πρέπει να ενισχύσουμε του μηχανισμού συνεργασία σε μεθοριακό επίπεδο ανάμεσα στα, στη θεσμική συνεργασία, την επίσημη α πούμε, αλλά πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μα και τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση κατά την εκπόνηση των ε, πολιτικών. Στα πλαίσια μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Θα πρέπει επίση να υπάρχει απόλυτη γνώση ε, της κατάστασης των, προβληματικών, των, των προβλημάτων ε, από τις τοπικές και αρχ, άλλες αρχές. Τα προγράμματα συνεργασίας ε, διεύρυναν την οικονομία που βασίζεται στη γνώση σε όλη την ε, Ένωση, το η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεγαλύτερη έρευνα, μεγαλύτερη ανάπτυξη και με αυτόν τον τρόπο θα τονώνουμε και τις ε, επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπάρχει μια διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας. Βελτίωσαν την πρόσβαση μεταξύ των συνόρων, την κοινή διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος. Λείπει όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ε, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει πραγματικά μια ευρωπαϊκή θεώρηση ε, υπό την ε, ε, ευγενική έννοια του όρου. Ε, το θέμα της μετανάστευσης. Ε, περιμένω να δω κάτι σχετικά με τη μετανάστευση και μέσα στην έκθεση. Ως μια, δηλαδή, ως ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της α, μετανάστευσης. Ο κύριος Ροπέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μ' αρέσει αυτή η έκθεση. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει όντως. Θα ήταν λάθος να σκεφτούμε το αντίθετο. Ε, τα περισσότερα κρατημέλη σήμερα έχουν πλήρως ανεπτυγμένες περιφερειακές πολιτικές και κρατική πολιτική που καλύπτει διάφορες επιμέρους περιοχές. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπως η δική μου που δεν έχουν ε, χωριστό σχεδιασμό αναπεριφέρειες. Δηλαδή, σχεδιάζουμε σε επίπεδο χώρας. Υπάρχουν διάφορες, ε, διαφορές λοιπόν από χώρα σε χώρα και δεν υπάρχει ένας και μόνο μηχανισμός για να απεικονίζει και να ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορές. Εμείς ε, στη φάση του σχεδιασμού καλύπτουμε όλη τη χώρα και αυτό δεν είναι φυσικά σωστό. Ε, Σχεδιάζοντα τι περιφερειακέ πολιτικέ, λοιπόν, τα κρατη θα πρέπει να το λάβουν υπόψη αυτά αυτέ τι διαφορέ δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τι ε, μεθοριακέ περιοχέ, συνήθω σκεφτόμαστε την όμορη χώρα. Εγώ ζω πολύ κοντά στην ε, Λευκορωσία, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα ζω. Η χώρα αυτή ε, δεν είναι και πολύ και παράδειγμα και πρότυπο δημοκρατίας και ανάπτυξης. Εν τη αυτή περιπτώση καταλαβαίνετε τα επιπρόσθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Φερρυπίν. Εκείνοι που εξαρτώνται, ας πούμε, ξέρετε ότι δεν διαλέγει κανένα τους γειτονές του και μερικές φορές εξαρτώμαστε από τους γειτονές μας. Ε, οι περιφέρειες ας πούμε, που έχουν σύνορα με λιγότερο δημοκρατική ανάπτυξη ή με χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο είναι συνήθως σε δυσκολότερη θέση. Οι περιφέρειες αυτές ε, είναι συνήθως απομακρυσμένες από τα κέντρα, έχουν ε, πιο πτωχές και ανεπαρκείς υποδομές και ο κόσμος αγωνιά για το μέλλον του. Όταν μιλάμε λοιπόν για την περιφερειακή πολιτική, θα πρέπει να σκεφτόμαστε εάν ο κόσμος θέλει να ζει σε αυτές τις περιοχές. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Πρέπει να αξιολογήσουμε λοιπόν την περιφερειακή διάσταση και να σκεφτούμε Πώς θα εξαλείψουμε αυτές τις διαφορές. Επίσης, υπάρχουν προβλήματα που είναι χαρακτηριστικά όχι μόνο της, που είναι χαρακτηριστικά όχι της χώρας, αλλά του γείτονα. Η Λευκορωσία ε, φτιάχνει ένα νέο πυρηνικό σταθμό, ας πούμε, ένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ το τοπικό επίπεδο, τον τοπικό πληθυσμό, σε διάφορα επίπεδα. Αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο θεωρείται μη ασφαλές εργοστάσιο. Θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και για μας, τους λετονούς. Θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι κανόνε, α πούμε, τόσο ώστε να δημιουργούν κάποια αναχώματα και να υπάρχουν κανόνε για το πώ μπορεί να ε, συμπεριφέρεται μια γειτονική χώρα. Και καλό θα ήταν, α πούμε, ειδικά όταν θέλει κάποιο να χτίσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο ή να χτίσει κάτι άλλο, α πούμε, να διαπραγματευόμαστε λιγάκι. Γιατί αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα, πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Έρμο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, και ε, ε, εγώ προέρχομαι από μια περιοχή που συνορεύει με Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία κατ' χώρες. Όποιος λοιπόν θέλει να μάθει πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει μια πενταετή, πενταάμινη πρακτική στο γραφείο μου σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Πρόκειται για προβλήματα αναγνώρισης διπλωμάτων πτυχίων σχετικά με την παροχή συντάξεων τις, ε, τα επιδόματα υγείας, αναπηρίας. Ε, είναι μια τεράστια λίστα προβλημάτων τα οποία συνεχίζουν να ε, υπάρχουν σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για αυτό. Δύο θέματα τώρα για την ανακοίνωση της Επιτροπής. Χαίρομαι ιδιαίτερως για το ότι το έκανε αυτό η Επιτροπή. Και ε, φυσικά με αυτό τον τρόπο, βέβαια δεν ανακαλύπτει ξαφνικά η Επιτροπή έτσι την ε, σημασία των παραμεθόριων περιοχών, όμως ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να αφιερώσουμε τον χρόνο ε, ώστε να βρούμε τις καλύτερες απαντήσεις. Υπάρχουν, προ, υπάρχουν προβλήματα διότι δεν γνωρίζουμε ποια νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί. Η μία ή η άλλη, πολύ συχνά όμως κανένα κράτος δεν θέλει πραγματικά να να λάβει την ευθύνη για το πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο εμείς όταν μιλάμε για προβλήματα θα πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι πιο καινοτόμα και όταν ε, είναι ένα, τόσο, ένα τέτοιο ε, πρόβλημα όπως είναι για την αναγνώριση κάποιων πτυχίων ε, τότε να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή ε, το οποίο στη συνέχεια στην άλλη περιοχή της αντίστοιχης χώρας θα ε, ισχύει. Και ένα άλλο ε, θέμα το οποίο πρέπει να συμπεριλάβουμε είναι ότι τα χρήματα τα οποία επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε προγράμματα Interreg και το τελευταίο σεντ θα πρέπει να ε, επενδύεται ορθά διότι αυτά τα προγράμματα αποτελούν μια ε, βάση ε, για να λυθούν τα προβλήματα αλλά ταυτόχρονα και να ταυτοποιήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και όταν αναγνωρίσουμε την ύπαρξη αυτών σε μια περιοχή τότε ίσως να υπάρχουν και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν μια παράκληση προς την Κομισιόν αλλά και οποιονδήποτε άλλο ασχολείται με τις περιοχές, παραμεθόριες περιοχές Παρακαλώ επενδύσετε περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα, ιδιαίτερο όσον αφορά ε, τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό, να μην περιοριστούν οι δαπάνες, αλλά αντιθέτως να αυξηθούν παρακαλώ επίσης ε, απλουστεύστε τις όλες ε, διαδικασίες. Η ε, συνεργασία είναι κάτι υπέροχο που θέλει να υπογράψει ο καθένας, αλλά αν ελέγχεται 4-6 φορές το χρόνο λόγω διαχείρισης προϋπολογισμών, εν τέλει δεν έχει καμία όρεξη να ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αμαρούση. Δύο λόγια. Κανονικά η Μαρτίνα Άντερσον ε, έπρεπε να είναι εδώ για να ε, σχολιάσει αυτό το θέμα και θα αναφερόταν στην Ιρλανδία και στις συνέπειες του Brexit ε, για την Ιρλανδία. Και φυσικά, μιλώντας για το θέμα των μεθοριακών περιοχών, δεν μπορούμε να ξεχνούμε το θέμα του Brexit. Και μάλιστα συναντήθηκα με πρόσωπο της Μεγάλη Βρετανία που βρέθηκε στι Βρυξέλλε και μα είπε ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα συνεργασία μεταξύ γαλλικών περιοχών και βρετανικών και διαρωτώνται οι περιφέρειες αυτέ οι περιοχές αυτέ. ποιο θα είναι το μέλλον αυτών των ε, προγραμμάτων συνεργασία. Οπότε καλό θα ήταν να εγκύψει αυτό το θέμα ο εισηγητή μα, παρόλο που γνωρίζουμε ότι εκρεμούν οι διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να περιπλέκουμε ή να κάνουμε δύσκολο τη ζωή του Επιτρόπου Μπαρνιέ, που είναι επικεφαλή των διαπραγματεύσεων. Και α μην ξεχνούμε και τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ που έχουν ακόμη μεγαλύτερε ιδιαιτερότητε. Συνήθω είναι απόμακρα νησιά, δεν έχουν καν χερσαία σύνορα και είναι πολύ ιδιάζουσα η δική του θέση. Γι' αυτό και θα καταθέσω τροπολογίε, ειδικά για, το, για την προβληματική των εξόχω απόκεντρων περιοχών και δι των νησιωτικών. Ο κύριος Βανίλ Mm. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είκοσι πέντε χρόνια διασυνοριακής ε, συνεργασίας έχουν περάσει και για ποιο λόγο λοιπόν ε, ξαφνικά ε, παρατηρούμε ότι δεν είμαστε παγκόσμιος πρωτοπόρος πάνω σε αυτό. Ε, για ποιο λόγο λοιπόν συνεχίζουν να υπάρχουν τόσο πολλά εμπόδια. Τα εργαλεία τα οποία έχουμε ε, είναι αναποτελεσματικά. Ε, για, εφόσον αυτό είναι ο λεφτό στο δωμάτιο, για ποιο λόγο δεν μιλάμε για όλο αυτό. θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην προηγούμενη περίοδο αλλά και στην τωρινή. Ε, είχαμε μια, είχαμε μια ομάδα ε, εδαφικής συνεργασίας. Έχουμε ε, περιοχές που βρίσκονται 100-150 χιλιόμετρα από τα σύνορα και υπάρχει η δυνατότητα να συνεργαστούν σε ζητήματα τα οποία αφορούν για παράδειγμα την αγορά εργασίας για να υποφεληθούν από την οικονομία κλίμακας. Αυτό θα, για να εφαρμοστεί θα πρέπει να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι περιοχές να εργάζονται πάνω σε αυτό. Αυτό δεν αφορά όλες τις περιοχές, μονάχα αυτές κοντά στα σύνορα ε, και είναι ξεκάθαρο λοιπόν ποιες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν ε, και σε ποιου τομεί για τις ε, μετακινήσεις, μεταφορές, εργασίας, παροχή υπηρεσιών ε, θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν επίσης ε, να μας πει που ε, πρότειναν αυτό το 2% για να βελτιωθεί η κατάσταση. Όμως άμα συνεχίσουμε με αυτή την ίδια πορεία όπως κάναμε και τα τελευταία 25 χρόνια, ναι είναι καλή διαφήμιση όμως τίποτα παραπάνω. Αν λοιπόν εξετάσουμε την κατάσταση από τη σκοπιά του ε, Brexit, την ε, προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στη Βόρεια Ιρλανδία και είχαμε ε, τη δυνατότητα να δούμε ότι τα εργαλεία τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας εκμεταλλεύονται, τα εκμεταλλεύονται ιδιαίτερως χάρη στο Interreg και αυτό σημαίνει ότι ότι τα σύνορα ε, παίζουν πολύ, ε, σε πολύ σημαντικό ρόλο, όμως τώρα ξαφνικά εισάγονται ε, σύνορα μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας. Το Κοινοβούλιο βέβαια δεν χαίρεται ιδιαίτερως γι' αυτό, δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις πάνω σε αυτό, όμως με βάση τις συζητήσεις που έχουμε μέχρι στιγμής, ίσως θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε την ευθύνη πάνω σε αυτό και να δούμε τις περιοχές εκεί, αυτό ίσως να ήταν ένα εργαλείο το οποίο θα απέφερε αποτελέσματα και υπάρχει στο πλαίσιο της παρούσας νομοθεσίας. Οπότε λοιπόν ε, μπράβο στην Κομισιόν για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση και ε, στον ε, εισηγητή. Όμως ε, πού βλέπετε να συνεχίζεται αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε ως την επόμενη αξιολόγηση για να δούμε ότι δεν κάναμε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ επιγραμματική. Η ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών ε, είναι αξιέπαινος στόχος. Ε, και γενικά η διακριτική συνεργασία είναι απρόσκοπτη, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της διαπεριφερειακής συνεργασίας ε, σε σχέση με την Ανατολική Σλοβακία και έχουμε ένα σύντομο χερσαίο σύνορο με την Ουκρανία 100 χιλιόμετρων και εκεί υπάρχει πρόβλημα συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ σκοπεύει να αντιμετωπίσει στο μέλλον τέτοια προβλήματα δυστοκίας σε περίπτωση διαπεριφερειακής συνεργασία, γιατί η Ουκρανία είναι σημαντικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν ώψη της, της μα μας έχουμε επενδύσει ε, πολλά κονδύλια εκεί. Διαπιστώσαμε όμω ότι τελευταία έχει ανασταλεί η χρηματοδότηση ε, πέντε διασυνοριακών σημείων διέλευσης ε, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβακία γιατί δεν πληρούσαν υποτίθεται τις ε, απαραίτητες προϋποθέσεις. Και είχαμε και το κονδύλιο προς την Ουκρανία. Οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία Σλοβακίας και Ουκρανίας είναι απαράδεκτες. Πλησιάζει και το Πάσχα και αν θέλετε κάντε μια βόλτα στην Σλοβακία, στα σύνορα με την Ουκρανία, θα χρειαστείτε πολλή ώρα για να περάσετε τα σύνορα. Είναι απαράδεκτες συνθήκες και η τοπική αυτοδιοίκηση στις παραμεθόριες περιοχές δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην τεράστια ζήτηση. Γι' αυτό και είναι πολύ χρονοβόρες διαδικασίες διέλευση των σύνορων. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ενθαρρύνει την Ουκρανία για να βελτιώσει την κατάσταση για τη δική τη πλευρά των σύνορων και πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η διασύνοριακή συνεργασία. Αλλά έχουμε πε... περιοχές που έχουν εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί από μόνες τους χώρες δεν μπορούν να επιλύσουν προβλήματα διασυνοριακής συνεργασίας. Θα πρέπει να τους βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Όλμπριχτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το θέμα του προηγούμενου πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου ε, και το πρόγραμμα EGTC που με απασχόλησε γιατί ήμουν εισηγητής για το προηγούμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο του 2013. Και μετά από μια δεκαετία περίπου, όπως είπε ο κύριος Χέτμαν, δεν έχουμε προχωρήσει σχεδόν καθόλου. Η κατάσταση είναι η ίδια. Θα σας παρουσιάσω καταρχήν το πρόβλημα και θα κάνω και τρεις προτάσεις. Το πρόβλημα δεν οφείλεται στις ε, περιφέρειες, σε ευρύτερες περιφέρειες, αλλά στην έλλειψη συμπληρωματικότητας των νομικών συστημάτων ε, των χωρών μελών. Αν έχουμε δύο όμερε χώρες με διαφορετικά νομικά συστήματα, υπάρχει μια αναντιστοιχία. Οπότε δεν μπορούμε να αναπτύξουμε την, τη συμπληρωματικότητα. Γιατί ε, προσπαθήσαμε να προωθήσουμε την διαμεθοριακή συνεργασία για να βρούμε κάποιες έκτακτες λύσεις σε στι παραμεθόρειε περιοχέ, στι όμορε περιοχέ, για να αποφευθούν τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω τη αναντιστοιχία των νομικών καθεστώτων. Οπότε το ιδανικό θα ήταν το σύνολο του συστήματο να είναι συμπληρωματικό. Να είναι συμπληρωματικά τα νομικά καθεστώτα μεταξύ των χωρών. Αλλά δεν τα καταφέρουμε σε εθνικό επίπεδο, τουλάχιστον να, να το επιχειρήσουμε εκτάκτως σε περιφερειακό επίπεδο. Το πρόβλημα δεν οφείλεται ε, στα, στη Σλοβακική περιφέρεια που συνορεύει με την Πολωνική περιφέρεια. Το πρόβλημα ε, είναι σε κεντρικό επίπεδο μεταξύ της Σλοβακικής κυβέρνησης και της Πολωνικής κυβέρνησης. Και αυτό αντικατοπτρίζεται σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά υπάρχει σε εθνικό επίπεδο. Και μερικέ φορέ φτάνουμε σε ακραίε καταστάσεις πραγματικά λόγω αυτή τη έλλειψη πληρωματικότητα. Γι' αυτό ε, ας κοιτάξουμε τι λεπτομέρειε. Και τι λένε οι λεπτομέρειε. Τι μα είπε ο Λάμπερτ. Η Επιτροπή των Περιφερειών μας υποχρεώνει σε συνεχή παρακολούθηση του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας. Και η τελευταία ενημέρωση που μας έκανε η Επιτροπή των Περιφερειών ήταν ερώτηση τι λειτουργεί το σύστημα, θα πρέπει να αλλάξει μετά το 2020 ή όχι. Δεύτερον, υπάρχει μια διαφορά μετά, μετά από μια δεκαετία ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ε, συνόρων Σέγγεν και των συνόρων εκτό χώρου Σέγγεν. Ποια είναι η κατάσταση στα σύνορα μεταξύ χώρε εντό και εκτός Σέγγεν, γιατί υπάρχει το θέμα της ελεύθερη διακίνησης των προσώπων και ελεύθερη κυκλοφορία ε, των προϊόντων. Γιατί έχουμε την περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ε, έχουμε την ίδια κατάσταση με αυτή των χωρών Σέγγεν. Επίση, τι γίνεται με τι χώρε εντό και εκτό Ευρωζώνη. Παράδειγμα, Σλοβακία, στι α, περιοχέ. Υπάρχουν διαφορέ μεταξύ α, ε, χωρών μελών τη Ευρωζώνη και χωρών εκτός Ευρωζώνη. Θα πρέπει και αυτά να τα δούμε. Το θέμα δεν είναι αν θα αναπτύξουμε ή όχι τη διαπεριφερειακή συνεργασία, αλλά το πώ θα χρησιμοποιούμε του διάφορου μηχανισμού και θα του προσαρμόζουμε στι ιδιαιτερότητε τη κατάσταση. Και η λύση ε, είναι και περισσότερα κονδύλια διασυνοριακά γιατί ακόμη είναι πολύ χαμηλά τα κονδύλια. Θα πρέπει να ενισχυθούν. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία, αλλά για να υλοποιήσουμε την ενίσχυση θα πρέπει να γίνει πρώτα μία ανάλυση και λεπτομέρειε μεταξύ χωρών Σέγγεν και εκτό Σέγγεν, Ευρωζώνης και εκτό Ευρωζώνης, περιφερειακές και πιο κεντρικέ. Με διασυνοριακό φυσικά χαρακτήρα και διάσταση. Ευχαριστώ. Εγώ μπορώ να σας ε, διηγούμε ώρες ολόκληρες ιστορίες για σύνορα εντός και εκτός έγκεν και περιφέρειες ή ε, σύνορα και περιφέρειες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά σίγουρα είναι εύλογο όλα αυτά τα ερωτήματα. κύριος Χάουαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 25 χρόνια δεν είναι και μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενώ η ιδέα του κράτους έθνους υπάρχει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ε, και λογικό είναι που υπάρχει μια μεγάλη προσήλωση σε αυτό. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί συχνά οι φραγμοί που υπάρχουν ε, διασυνοριακά είναι πολιτιστικοί φραγμοί, όσο και οικονομικοί ή εμπορικοί ή νομοθετικοί. Ε, και πολλά από αυτά που μας είπαν αυτοί που επισκέφτηκαν την Ιρλανδία είναι ότι ο κόσμος ξέρει ότι η επανεμφάνιση των πολιτιστικών ε, φραγμών και επειδή υπάρχουν ε, διαφορετικές παραδόσεις θα δημιουργήσουν ε, τεράστια προβλήματα. Φυσικά οι Ιρλανδοί τα ξέρουν καλύτερα από μένα. Όμως, εκεί έχουμε σημειώσει μία τεράστια επιτυχία. Ο κύριος Βανίστερο και ο κύριος ε, το είδαν. Είδαν τι σημαίνει να εξαλείφεις κάποιους σημαντικούς μεθοριακούς φραγμούς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα Ιρλανδικά σύνορα είναι σε φανταστική κατάσταση. Υπάρχουν θέματα ε, αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων κτλ. Ε, και ένα βασικό θέμα για τις μελλοντικέ πολιτικές είναι αυτό που είπε ένα συνάδελφος. Να πούμε τι μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά η αμοιβαία αναγνώριση των α, επικοινωνιών, η προώθηση της, των πολιτικών αλλαγών και η αμοιβαία κατανόηση, η συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών αρχών ε, από τη μία και την άλλη μεριά των συνόρων. Τι πρόκειται. Αν, ας πούμε, αν βάλουμε περισσότερα λεφτά ε, στην ε, περιφερειακή πολιτική, αυτά τα λεφτά σε τι θα τα επενδύσουμε. Και τι θα, δώσει, και τι θα επιφέρει αυτό. Ε, τι θα δώσει τα περισσότερα πλεονεκτήματα στο εγγύς μέλλον. Ε, και το καλύτερο παράδειγμα εδώ είναι η Ιρλανδία, ας πούμε. Γιατί αν ε, σταματήσεις, ας πούμε, να, τον τοίχο, αν κατεδαφίσεις τον τοίχο, ας πούμε, θα έχεις πολλά ωφέλη. Ε, πριν από λίγα χρόνια πέρασα από το Κέντ, πήγαινα από το Κέντ, ας πούμε, στο Νοχ Παντουκαλέ. για ένα πρόβλημα υγείας, ε, για να το λύσω στην άλλη μεριά του καναλιού, ας πούμε. Ε, γιατί δεν μπορούσα, είχαμε προβλήματα στο Κέντ. Ελπίζω να συνεχιστεί. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι το χρόνο ε, 4 εκατομμύρια φορτηγά ε, περνάνε τα χερσαία σύνορα. είναι τεράστιο το θέμα αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ ψηλά αυτό το θέμα στην ε, ατζέντα του κυρίου Μπαρνιέ. Δεν θέλω να του περιπλέξω περιττό το βίο με αυτά τα θέματα. Αυτά ήταν τα σχόλια και οι προτάσει των σκιωδών εισηγητών και μελών τη Επιτροπή Ρέτζη. Και τώρα ο κύριο Φερέιρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο, να μα δώσει απαντήσει ενδεχομένω σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς όλα αυτά τα ερωτήματα. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που κάνει αυτή τη συζήτηση. Τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική. Επίκαιρη, πολύ συζήτηση. Ευχαριστώ τον κύριο Χέκμαν για την ανακοίνωση και περιμένουμε να δούμε και το κείμενο της, της ε, εκθεσής του. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω όλα τα και να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια από αυτά. Αυτά που ακούστηκαν περισσότερο. Ένα από τα ερωτήματα που είπαν πολλοί ευρωβουλευτές είναι τα θέματα τα οποία, ε, στα οποία εστιάζουμε. Ας πούμε, ορισμένοι λένε γιατί όχι μετανάστευση. Γιατί όχι περιβαλλοντική ε, πολιτική. Γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται. Ε, το πρόβλημα είναι συχνά σε εμπόδια λόγω συνόρων και σε διασυνοριακή συνεργασία που αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Άλλες είναι οι επιπτώσεις από σύνορο σε σύνορο αλλά υπάρχουν στους περισσότερους τομείς που μπορούμε να σκεφτούμε τα εμπόδια αυτά. Ίσως δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα, όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σύνορα με τη μία. Όπως είπε και σωστά η κυρία Νταμάτο, αυτή η ανακοίνωση προηγήθηκε από μία, μάλλον υπήρχε μία πρώτα μία πρώτερη τεράστια δημόσια διαβούλευση με ενδιαφέρομενους φορείς, με ακαδημαϊκούς, με πανεπιστημιακούς, για να εντοπίσουμε τα πιο συνήθη προβλήματα στη διασυνορική συνεργασία. Και από αυτή τη διαβούλευση, με την κοινωνία για τις διασυνοριακές περιοχές, εντοπίσαμε τα βασικά θέματα που εξετάζει η ανακοίνωση. Θεωρούμε ότι αυτά τα θέματα είναι αυτά όπου ζητάει ο κόσμος και οι περιφέρειες αυτές πιο συχνά να υπάρξει δράση. Εκεί όπου εστιάζονται περισσότερο τα προβλήματα, εκεί που εντοπίζονται περισσότερο οι δυσκολίες. Ο κύριος Χέτμαν έθεσε κυρίως τέσσερα ερωτήματα. Το πρώτο από αυτά αφορά αυτό που λέμε εμείς στο κεφάλαιο 3.2 της ανακοίνωσης, όπου η ανακοίνωση λέει ότι η εφαρμογή των ισχυουσών μεθόδων και εργαλείων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στην νομοθετική διαδικασία είναι σημαντικό να γίνει. Εκεί είναι η ενότητα όπου εξετάζουμε τα νομοθετικά θέματα στην ανακοίνωση. Το να ενσωματώσουμε τις μελέτες εδαφικών, αντικτύπου στην εσωτερική διαδικασία ε, μελετών αντικτύπου πριν υιοθετήσουμε νέα νομοθεσία. Αυτό που λέμε λέει, είναι τι, ότι οποτεδήποτε προτείνουμε ένα νέο νομοθέτημα μεγάλης εμβέλειας, στην προπαρασκευαστική φάση θα πρέπει να έχουμε μία μελέτη αντικτύπου και αυτό που ζητάμε, αυτό που θα θέλαμε, είναι το θέμα ε, της μελέτης αντικτύπου να εμπλουτιστεί, η μελέτη αυτή αντικτύπου να εμπλουτιστεί, ούτω ώστε να ασχολούμαστε εξειδικευμένα με τη συγκεκριμένη περιοχή στη μελέτη αντικτύπου και οι επιπτώσεις στις διασυνοριακές ε, περιοχές αυτές να εξεταστούν πολύ συγκεκριμένα πριν περάσει αυτό το νομοθέτη, νομοθέτημα. Γιατί όπως υπόθηκε, συχνά τα προβλήματα προέρχονται από την έλλειψη συνέπειας ανάμεσα στα διάφορα νομικά πλαίσια. Δηλαδή, ανάγκη να αξιολογήσουμε την επίπτωση που έχει στην περιοχή αυτή εκ των προτέρων είναι πάρα πολύ σημαντική. Δύο συγκεκριμένα ερωτήματα τέθηκαν επίσης. Ε, τα πιλωτικά προγράμματα και η προκήρυξη υποβολής πιλωτικών προγραμμάτων, αυτό έχει ξεκινήσει ήδη έχει ανοίξει η διαδικασία αυτή και καλούμε όλα τα κράτη-μέλη να στείλουν τις πληροφορίες αυτές. Ή μάλλον ε, καλούμε τους βουλευτές να στείλουν τις πληροφορίες στα κράτη-μέλη τους. Αυτή η προκήρυξη υποβολής προσφορών μιλάει για πιλωτικά project για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα, εντοπισμένα προβλήματα στα σύνορα, στα, στη Μεθόριο. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα πιλωτικά ε, για να δείξουμε ότι με το να εμπλέκουμε διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς ε, σε μια πολυεπίπεδη συμμετοχή μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Επίσης, αναφέρθηκε η ανάγκη για τις ε, ελίπουσες, τους ελείποντες κρίκους της αλυσίδας. Αυτή η μελέτη έχει οριστικοποιηθεί. Έχουμε λάβει την τελική εκδοχή την περασμένη εβδομάδα και στη μελέτη, στη μελέτη αυτή θα σας τη δώσουμε μετά τα απαραίτητα τεχνικά και διοικητικά βήματα που πρέπει να, από τα οποία πρέπει να περάσει. οργανώνουμε και ένα εργαστήρι ειδικό για αυτή τη μελέτη ε, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα περιφερειών και πόλεων. Διάφορες ερωτήσεις ακούστηκαν και τα EGTC, ε, την, τις ε, Ευρωπαϊκές Ομάδες Ενταφικής Συνεργασίας. Μήπως δεν αρκούν. Αρκούν, πρέπει να τις αναθεωρήσουμε. Μήπως τα κράτη-μέλη δεν τις χρησιμοποιούν. Οι ομάδες αυτές είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να επιληθούν πολλά προβλήματα σε διάφορα σύνορα. Η χρήση όμως εξαρτάται από τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν ε, δώσει το νομοθετικό πλαίσιο για να δημιουργηθεί αυτό το εργαλείο, υπό το οποίο οι εθνικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να κινητοποιηθούν για να, και να το χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να λύσουν τα προβλήματά του. Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Ε, η Επιτροπή των Περιφερειών μας είπε ότι η χρήση αυτών των ομάδων αυξάνεται σε διάφορες περιοχές. Και τώρα έχουμε τέτοιες ομάδες σε πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια που συνεργάζονται μέσω της χρήσης αυτών των εδαφικών ομάδων. Έχουμε επίσης ένα μεγάλο νοσοκομείο στα σύνορα μεταξύ Ισπανία και Γαλλία που χτίστηκε ως τέτοια ομάδα, ας πούμε, για να εξυπηρετήσει το, τον πληθυσμό και από τα δύο, τις δύο μεριές των συνόρων. Αρκεί, πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ένας από τους τομείς ε, που θίγει η ανακοίνωση είναι η συνέχεια που πρέπει να δοθεί στο εργαλείο που προτείνουν διάφορα κράτη-μέλη υπό την ε, πρώτη μάλλον υπό Ξεμβουργικής ε, Προεδρίας, η Ευρωπαϊκή Διασυνοριακή Σύμβαση. Αυτή η σύμβαση ήταν μια πρόταση από τα κράτη-μέλη, όπως είπα. Και πήγαινε προς την κατεύθυνση που είπε, νομίζω, ο κύριος Όλμπριχτ. Νομίζω ότι δηλαδή θα πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε τους κανόνες για να εναρμονίσουμε να εναρμονίσουμε τα όσα κάνουμε σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτή η σύμβαση θα δημιουργήσει και ένα νομικό πλαίσιο που θα μας επιτρέπει, θα επιτρέπει στις περιφέρειες των κρατών μελών να διαπραγματεύονται λύσεις μέσω των οποίων εναρμονίζουν τους κανόνες για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επίσης. Διάφορα σχόλια επίσης έγιναν για τα εξωτερικά σύνορα. Για τις ε, υπερπόντιες, υπερπεριφερειακές μάλλον περιοχές, μήπως ξεχάσαμε λοιπά. Όχι, δεν τα έχουμε ξεχάσει αυτά τα σύνορα, τα εξωτερικά. Απλώς έχουν διαφορετικά προβλήματα. Αυτή η ανακοίνωση δεν αντιμετωπίζει τα εξωτερικά σύνορα. Δεν αντιμετωπίζει τα θαλάσσια σύνορα. Δεν αφορά τις υπερπεριφερειακές και υπερπόντιες περιοχές. Γιατί έχουν τελείως διαφορετικά προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν προβλήματα αυτά σύνορα. Έχουν. Αλλά έχουν διαφορετικής φύσης προβλήματα. Κύριος Βανίστελ Ρόι τα είπε πολύ σωστά. Και μας ρώτησε γιατί έχουμε πρόβλημα. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι ρώτησε γιατί έχουμε πρόβλημα. Με όλα τα εργαλεία που έχουμε δημιουργήσει θα έπρεπε να έχουμε ακόμα προβλήματα στις εσωτερικά σύνορα. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση εστιάζει ακριβώς αυτό το θέμα. Σε αυτά τα προβλήματα που είναι επίμονα. Ενώ θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι θα έπρεπε να έχουν επιληθεί μέχρι τώρα. δεν έχουν επιληθεί πλήρω. Οι μελέτες που αναφέρει, στις οποίες παραπέμπει η ανακοίνωση Μιλάει, μιλάνε για τις πιθανές επιπτώσεις στις, στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης στις μεθοριακές περιοχές. Τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον, κυρίως. Σε αυτή τη συζήτηση αναφέρατε την ανάγκη να υπάρξει μια πολυεπίπεδη συμμετοχή. Να εμπλακούν οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς. Μπορούμε να δώσουμε τα εργαλεία, γιατί θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να συμμετάσχουν. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για αυτή τη συζήτηση. Είναι πολύ επίκαιρη, τη χρειαζόμαστε πραγματικά. Και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας για να συνεχίσουμε τη συζήτηση υπό οποιαδήποτε μορφή θέλετε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. Hetman, you have the floor. ευχαριστούμε ο εισηγητής μας ο κύριος Χέτμαν για να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πολύ λακωνικά. Στο τέλος ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τους συναδέλφους για την ιδιαίτερο ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψε. Ε, φαίνεται ότι συμπίπτουν οι απόψεις μας ό,τι φορά την ε, διάγνωση του προβλήματος και την ε, ανάλυση των ε, λύσεων που χρειάζονται δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων και των διαφορών στις παραδόσεις και στα πολιτιστικά θέματα. Αλλά αυτό που θέλουμε όλοι και είναι ο κοινός μας παρανομαστής είναι να διευκολύνουμε την καθημερινότητα 150 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που διαβιούν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια στις παραμεθόριες περιοχές. Και χαίρομαι ιδιαίτερος και θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκύπτει στα καθημερινά προβλήματα των ε, κατοίκων αυτών των περιοχών. Αυτοί που κάνουν, για παράδειγμα, έχουν εφρική ανεπάρκεια ε, και έχουν πρόβλημα στην, στις προσβάσεις της ε, υπηρεσίας υγείας, στην οικονομική περίθαλψη, στις υπηρεσίες παιδείας και σε διάφορα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους. Επίσης, αναφέρθηκε η πρόταση ενίσχυση των χρηματοδοτικών κονδυλίων ε, για τα διασυνοριακά προγράμματα μετά το 2020. Αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία του προγράμματος Interreg, της πρωτοβουλίας Interreg, γιατί πρόκειται για ειδικά προγράμματα και η έγκριση και δρομολόγηση εφαρμογή τους ε, προσκρούει σε πολλές δυσκολίες, πολύ περισσότερες από τις δυσκολίες που χαρακτηρίζουν άλλα προγράμματα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την επιπλέον γραφειοκρατική διατύπωση θα πρέπει να τη διορθώσουμε. Και μια και μιλούμε για την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, φανταστείτε όσοι είχαν την ευκαιρία να ε, εφαρμόσουν τέτοια προγράμματα έχουν πολύ ενδιαφέρουσες ε, εμπειρίες και μάλιστα μερικέ φορέ έχουμε δύο εταίρου ε, στι δύο πλευρέ των συνόρων, Μερικέ φορέ έχουμε και τρει εταίρου από τρει διαφορετικέ χώρε όμορε, οπότε θα πρέπει να έχουμε διευκόλυνση των συστημάτων για την προκήρυξη των δημόσιων διαγωνισμών, για τι προμήθειε και κατά την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αυτόν των περιοχών και θα πρέπει να διευκολύνουμε και σε διοικητικό γραφειοκρατικό επίπεδο την απλούστευση και θα πρέπει να διευκολύνουμε τη διασύνοριακή συνεργασία. Δεν θα αναφερθώ στην διασυνοριακή συνεργασία με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτή είναι διασυνοριακή συνεργασία σε εξωτερικά σύνορα. Και εγώ μένω σε τέτοια περιφέρεια και έχουμε γειτονικέ χώρε στην Ουκρανία και την Λευκορωσία. Αλλά εγώ δεν αναφέρθηκα σε τέτοιε περιπτώσει, γιατί δεν είναι αυτό το περιεχόμενο ούτε της εκθεσής μου ούτε της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι άλλο θέμα για μεταγενέστερη συζήτηση. Πάντως δύο είναι τα σημεία κλειδιά ε, και τα επισήμενα ο κύριος Βενίστερο. Ε, θα πρέπει καταρχήν ε, να, άρουμε, να δρήσουμε κάποια συμπεράσματα από την 25χρονη εφαρμογή αυτής της συνεργασία. συνεργασίας και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να βελτιώσουμε ποιοτικά την καθημερινότητα των κατοίκων των παραμεθόριων περιοχών. Και για να το κάνουμε θα πρέπει πρώτα να κλείσουμε τα σωστά διδάγματα από αυτή την 25χρονη μέχρι τώρα εφαρμογή για να προχωρήσουμε. Και πολύ σημαντικό είναι και εύστοχο αυτό που είπε ο κύριο Όλμπριχτ, ότι τα προβλήματα αυτά που ε, βασανίζουν τις ε, παραμεθόριες και διασυνοριακές περιοχές δεν είναι όλα τα ίδια. Γιατί μια εναρμόνιση ενδεχομένω των διατάξεων ε, δεν μπορεί να γίνει ούτε σε τοπικό ούτε σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται μεγαλύτερη εμπλοκή των κρατών μελών και αντίληψη των ε, ιδιαιτεροτήτων των ε, και των προβλημάτων των περιοχών αυτών, γιατί επαναλαμβάνω δεν υπάρχει ένα καλούπι για όλες. Ευχαριστώ. Περιμένουμε το σχέδιο έκθεσή σας για το Μάιο, κύριε Χέτμαν, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε και να αναλύσουμε τα προβλήματα της διασυνοριακής και της παραμεθόριας συνεργασίας. Αυτά. Ολοκληρώσαμε την απογευματινή μας ημερήσια διάταξη και να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα γίνει απεργία, έχει ανακοινωθεί απεργία των οδηγών ταξί και μην ξεχνάτε ότι στις 9 έχουμε ψηφοφορίες, γι' αυτό προγραμματίστε τη μέρα σας ώστε να έρθετε εγκαίρως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ολοκληρώνουμε το δημόσιο τμήμα της συνεδρίασής μας και θα ήθελα να ρωτήσω τους συντονιστές αν μπορούμε να περάσουμε αμέσως στη συνεδρία των συντονιστών που είχε προβλεφθεί για αργότερα λίγο. Ωραία, είναι παρόντες οι συντονιστές, οπότε θα αρχίσουμε αμέσω με τι συνεδρίες των συντονιστών και παρακαλώ όσοι δεν δικαιούνται να είναι παρόντες να αποχωρήσουν.